Queridos compañeros y compañeras, me toca. Αγαπητοί συνάδελφοι, έλεγχε σε μένα η τιμή της έναρξης της σημερινής συνεδρίασης. Θα κάνω μια ενημέρωση και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρουμπίχ που είναι ορμόδιο για την ακρόαση με θέμα του νέου επιχειρηματίε και θα προεδρεύσει σε αυτήν. Έχουμε πρώτο σημείο της σημερινής διάταξης, την έγκρισή τη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σχόλια για το θέμα αυτό. Αν όχι, περνάμε στο δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης, της ανακοινώσης του Πρόεδρου. Έχετε τις, έχουμε όλες τις γλώσσες για διερμηνία. Και μην ξεχνάτε ότι η συνεδρίασή μας αναμεταδίδεται και με webstream. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ρούμπιχ, να καλωσορίσω μία ομάδα του ε, Γερμανικού Συμβουλίου Φεντεραλιστών από τη Γερμανία. Καλώς ήρθατε. Φαντάζομαι θα ενδιαφέρεστε για το σημερινό θέμα των ε, νέων επιχειρηματιών και είναι φοβερή σύμπτωση ότι σα φιλοξενούμε την ημέρα ακριβώ που έχουμε την ακρόαση με θέμα του νέου επιχειρηματίες. Αυτά και περνάμε στο πρώτο σημαντικό θέμα της ημερήσια διάταξης που είναι η ακρόαση με θέμα το έρασμο για του νέου επιχειρηματίε. Έχετε το λόγο κύριε Ρουμπίχ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι για μα όλου είναι μεγάλη χαρά το ότι εδώ σήμερα έχουμε διοργανώσει αυτό το, αυτή την ακρόαση με θέμα Εράσμους για νέους επιχειρηματίες. Το πρόγραμμα για μας στο ε, Κοινοβούλιο, δεδομένης και της ε, ανεργίας που επικρατεί στην νεολαία, είναι μεγάλης προτεραιότητας. Ω πλωτικό πρόγραμμα ξεκίνησε από το στο Κοινοβούλιο το 2008 και έκτοτε έχει στεφθεί με επιτυχία το πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο Πιτέλα, ο οποίος ενεργά συμμετείχε στην όλη διαδικασία. Και κυρίως χαίρομαι που καλωσορίζω εδώ τον συνάδελφο Κρόιτσμαν, ο οποίος ως εισηγητής φρόντισε για την διαμορφώση του προγράμματος και θα ήθελα κατευθείαν να τόσο το λόγο λοιπόν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, ο κύριος Κρόιτσμαν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι και επισκέπτε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση εδώ πέρα στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Με μεγάλη μου χαρά να σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία για το πρόγραμμα Εράσμους για Νέες επιχειρηματίες. Ε, εγώ ω εισηγητής τα θεωρώ σημαντικά τα στοιχεία αυτή. Καταρχάς, ε, να σα μιλήσω για τις ε, θέματα ανταγωνιστικότητας για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις σχετικές επιδοτήσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως είπα. 20 Ιουνίου, στα πλαίσια του τριμερούς ε, διαλόγου, πετύχαμε μόλις ε, συμφωνία με το Συμβούλιο. Χαίρομαι γιατί πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σημαντικό για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση στην Ευρώπη και ιδιαίτερω σε περίοδους κρίση, όπου πραγματικά η οικονομική κατάσταση έχει συρρυκνωθεί σε όλε τι χώρε, ο ρόλος ε, της ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων πραγματικά είναι ύψης της σημασίας. Εμείς ε, πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για το μοναδικό πρόγραμμα που πραγματικά απευθύνεται σε αυτές τις εταιρείες, το πρόγραμμα Κόσμο, με συγκεκριμένα μέτρα για την μείωση της γραφειοκρατίας, για την επιδότηση και την προώθηση της επιχειρηματικότητας. χρηματοδοτείται από τη χρηματοδοτική περίοδο 2014 με 2020 και να σας πω ότι στην αρχή είχαμε προτείνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0,3 δισεκατομμύρια, αλλά δυστυχώς έγιναν περικοπές ε, στη λάθος, στο λάθος κλάδο. Και έτσι το πρόγραμμα COSME ε, ε, μειώθηκε λίγο σε ό,τι αφορά τα κονδύλια. Σε ό,τι αφορά την προώθηση της επιχειρηματικότητας, σημαντικό είναι τα προγράμματα κινητικότητας για νέους επιχειρηματίες και για την τεχνογνωσία των νέων, προκειμένου να αναπτύξουν ικανότητες και να αναπτύξουν τις ικανότητες τους σε ό,τι αφορά θέματα τεχνολογίας. Τι εννοείται, Εννοείται ασφαλώ το Εράσμο για νέου επιχειρηματίε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε ωστόσο να χρησιμοποιηθεί μια πιο γενική διατύπωση προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία σε τα επόμενα 7 χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα εξασφάλισε και μα καθησύχασε ότι σε, κά... καμία περίπτωση δεν πρόκειται να διακοπεί το πρόγραμμα Εράσμου για νέου επιχειρηματίε. Χαίρομαι λοιπόν που τα πληθυκά αυτά προγράμματα συνεχίζονται και μπορούν να εφαρμοστούν για ακόμα 7 χρόνια. Το Εράσμος για νέες επιχειρηματίες δημιουργήθηκε το 2009 και όπως είπε ο συνάδελφος Ρούμπιχ αποδείχθηκε μια ιστορία επιτυχέστατη. Έχουν γίνει υποδεκτές 204 αιτήσει από νέους επιχειρηματίες. Πρόκειται για μια κατάσταση διπλού ωφέλους ανταλλαγής ε, εμπειριών, διεύρυνσης των οριζόντων. Τι αναφέρεται στο πρόγραμμα του κόσμου, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μπορεί έτσι να εφαρμόζει τα προγράμματα κινητικότητας για τους νέους. Και αυτό ε, από το απόσπασμα της έκθεσης του Δ. Ρούμπιχ. Η Ευρωπαϊκή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε να ε, ήταν υποχρεωμένη να τα εφαρμόσει αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώ αυτό δεν έγινε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν στην επόμενη προγραμματική περίοδο θέλει να έχει ε, επαρκή ευελιξία για να είναι προετοιμασμένη για κάθε περίπτωση. Ο προπολογισμό για το κόσμο είναι στο 2,5% 2,5% του προπολογισμού των 2,0 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ε, θεωρούμε ότι μπορεί να αφιερώσει μεγαλύτερα κονδύλια στο κλάδο αυτό. Αν θέλει όμως ε, να αυξήσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει πράξεις κατά εξοδοσιοδότηση, στην οποία περίπτωση μπορεί να προβάλλει βέτο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ευέλικτη διαμόρφωση του κόσμου σημαίνει ότι εμεί Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τι αρμοδιότητε μας προκειμένου να αξιοποιηθούν και να εξαντληθούν οι δυνατότητε για χρηματοδότηση και να επαρκούν τα κονδύλια. Ιδιαίτερα σε περίοδους μεγάλης ανεργίας θα πρέπει να υποστηρίζουμε τέτοια προγράμματα και θα ήθελα να πω το εξή. Οι νέοι σήμερα έχουν μία ευκαιρία. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να είναι ανεξάρτητοι. Πάντα έχουμε προβλήματα όταν στη ΣΥΠΑ για παράδειγμα βλέπουμε ποια είναι τα αριθμητικά στοιχεία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκύπτει ότι στερούμε πάρα πολύ. Είναι μία τεράστια ευκαιρία. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά μας κατηγορούν ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά από τον πολίτη. Αν θέλουμε λοιπόν να προσεγγίσουμε τον πολίτη, ακριβώς με αυτά τα προγράμματα χρηματοδότησης μπορούμε να τον προσεγγίσουμε. Από εκεί, από αυτά τα προγράμματα θα προκύψουν θετικά αποτελέσματα και θα βελτιωθούν οι καταστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει στην Αβλεφερούμπιχ να φροντίσουμε να μην ε, περικοπεί υπερβολικά το πρόγραμμα. Αντιθέτως, μήπως μπορεί να επεκταθεί η χρηματοδότησή του παρά τις ε, χαλεπούς καιρούς που ζούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε Κρόιτσμαν. Λέει ο κύριος είχε να αναφέρω ότι ασφαλώς πρόκειται για δημόσια ακρόαση και βρισκόμαστε, μεταδιδόμαστε και στο διαδίκτυο. Να παρακαλέσω τους ε, συναδέλφους, όλους τους ομιλητές, να μιλούν τη γλώσσα τους, εφόσον αυτό είναι δυνατόν. Έχουμε και το φάκελο για το σχετικό πρόγραμμα και έτσι περνάμε στον πρώτο προσκεκλημένο μας, τον κύριο Κρίστιαν Βάινμπεργκερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τη Γενική Διεύθυνση ε, Επιχειρήσεων. Ήταν ένα από, από τους παράγοντε παράγοντες ε, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την προώθηση του προγράμματος αυτό. Πάντα υποστήριζε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν τον ευχαριστώ ιδιαίτερος και του δίνω το λόγο. Thank you very much, Mr. Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να σας ενημερώσω πέντε χρόνια μετά την έναρξη της πρώτης πιλωτικής δραστηριότητα για την επιτυχία του προγράμματος αυτού. Θα γνωρίζετε ότι το κόσμο είναι το δημοσιονομικό σκέλος, αλλά έχουμε και πολιτικό σκέλος για την επιχειρηματικότητα και τις δραστηριότητες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι το Small Business Act. Και το Εράσμος για τους νέους επιχειρηματίες ήταν ένας από τους άξονες που ήδη από το 2008 αναγγέλθηκε στο νομοσχέδιο για τις μικρές επιχειρήσεις και όταν ανέλαβε ο Αντιπρόεδρος Σταγιάννη ήρθε σχεδόν αμέσως ε, στο Στρασβούργο για να εκφράσει την υποστήριξή του για το πρόγραμμα ήδη από την αρχή της εφαρμογής του και εξακολουθεί να είναι ένθερμος υποστηρικτής του προγράμματος αυτό, Επιτρόπος Ταγιάννη. Όπως σας είπα, έχει το πρόγραμμα αυτό συγκεκριμένο ε, αντίκτυπο και απτά αποτελέσματα στους Ευρωπαίους πολίτες. Και αυτό προσπαθούμε να ενισχύσουμε και στο μέλλον. Θα ήθελα εν συντομία να αναφερθώ σε ορισμένα στοιχεία και κάποιες ανησυχίες στα πλαίσια του προγράμματος. Μια σύντομη εισαγωγή πρώτα για τον τρόπο λειτουργία του και κατόπιν ε, έχω μια διαφάνεια με τα αποτελέσματα, τους στόχους και φυσικά κάποια συμπεράσματα και για το τι μέλη γενέστε. Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει πρόθεση να διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών, ε, δικτύωση και ε, εκπαίδευση για νέους επιχειρηματίες ε, με πειράματα με ανάδοχους επιχειρηματίες ε, και νέους επιχειρηματίες. Ένας, ανάδοχος επιχειρηματίας, ένας νέος επιχειρηματίας ε, επιλέγει έναν ανάδοχο και περνά μαζί του ένα με έξι μήνες. Και σε αντίθεση με το πρόγραμμα για τους φοιτητές και σπουδαστές, το έρασμος για τους φοιτητές που όλοι γνωρίζετε, το έρασμος για τους νέους επιχειρηματίες δεν προβλέπει ασύμμετρη ανταλλαγή. Είναι συμμετρική ανταλλαγή εδώ. Είναι στο ίδιο επίπεδο, δηλαδή ο νέος και ο ανάδοχος ε, επιχειρηματίας που περνάει πέντε ώρες την εβδομάδα με τον νέο επιχειρηματία για να καταστήσει υποφελές το πρόγραμμα. Και μάλιστα έχουμε στην ακρόαση και, εκπροσω... έναν ανάδοχο επιχειρηματία και έναν νέο επιχειρηματία που θα μας παρουσιάσουν και εμπράκτος τις εμπειρίες τους. Θέλουμε υγιή startup, γιατί για μια υγιή επιχειρηματικότητα θέλουμε όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες να ξεκινήσουν επιτυχία την επιχείρησή τους. Όχι δηλαδή απλώς έχω μια ιδέα θα την εφαρμόσω, αλλά να συζητήσω με έναν πεπειραμένο επιχειρηματία για να βρω τον καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσω την επιχείρησή μου, ώστε να μειωθεί ε, το έπακρο το ποσοστό αποτυχίας. Αλλά το πρόγραμμα αυτό έχει πλεονεκτήματα και για τους αναδόχους επιχειρηματίες λόγω της διεθνοποίησης, γιατί ο νέος επιχειρηματής είναι από άλλη χώρα, αλλά και από άποψη καινοτομία. Γιατί οι νέοι επιχειρηματίες φέρνουν ένα φρέσκο μυαλό, μια φρέσκα, φρέσκια προοπτική και νέες ιδέες στον ανάδοχο επιχειρηματία που θα τον επιτρέψει να κατακτήσει νέες αγορές και να αναπτύξει νέα προγράμματα και υπηρεσίες. Οπότε στόχος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Η επόμενη διαφάνεια μας δείχνει κάποιες λεπτομέρειες για το σύστημα. Έχουμε τις ανταλλαγές μεταξύ των επιχειρηματιών, αναδόχων και νέων. Για να γίνουν εφικτές αυτές οι ανταλλαγές έχουμε και κάποιους ενδιάμεσους οργανισμούς, 150 προς το παρόν, που οργανώνουν αυτές τις ανταλλαγές. Οι λεπτομέρειες ε, των, του έργου τους ε, αργότερα. Τώρα, για τον νέο επιχειρηματία τα πλεονέκτηματα είναι ότι, ότι θα ε, λάβει συμβουλές και θα διδαχθεί από την εμπειρία του πιο έμπειρο επιχειρηματία, θα δημιουργήσει διεθνείς επαφές, δικτύωση, ε, γνώση για τις νέες αγορές, αλλά και κάποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τώρα για τον ανάδοχο επιχειρηματία, ίσως τα πλεονεκτήματα δεν είναι ορατά εξ αρχής, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν γιατί και οι ανάδοχοι επιχειρηματίες θα ενισχύσουν τις γνώσεις τους για τις διεθνείς αγορές, μπορούν και να βοηθήσουν κάποιον, μπορούν να βοηθούν να, να διεισδύσουν και σε διεθνείς αγορές και να δημιουργήσουν και εταιρικέ ε, σχέσεις. Γνωρίζουμε από την ε, έρευνα ότι 50% των επιχειρηματιών εξακολουθούν και μετά τις ανταλλαγές να διατηρούν ε, επαφές μεταξύ τους. Τώρα, πώς λειτουργεί το σύστημα. Πρώτο βήμα, αίτηση και των δύο επιχειρηματιών. Έχουμε εδώ τον ανάδοχο στη Γερμανία και τον επιχειρηματία στην Ισπανία. Έχουν online έγγραφο με το, το αιτιολογικό. Ε, εξετάζεται η αίτηση αυτή από τον ενδιάμεσο οργανισμό και εφόσον πληρούνται οι προποθέσει με την αυστηρότερη προπόθεση είναι το σοβαρό ενδιαφέρον για έναρξη επιχείρηση. Δεν αρκεί δηλαδή να σπιτήσει να πει είμαι άνεργο γιατί να μην γίνουν επιχειρηματίε, Εδώ μιλούμε για σοβαρούς ετούντε που θέλουν όντω να ανοίξουν μια επιχείρηση ή να την έχουν πρόσφατα ξεκινήσει. Εφόσον συντρέχουν όλε αυτές οι προποθέσει μέσω του μεσάζοντος οργανισμού έρχονται σε επαφή, ε, γίνονται δεκτέ αιτήσει. Τώρα γίνεται μια αναζήτηση και ένα συντέριασμα καταρχήν στις χώρες ενδιαφέροντος και αυτός ο ενδιάμεσος οργανισμός κάνει μια έρευνα και βρίσκει τους κατάλληλους ε, επιχειρηματίες, τους πιο ταιριαστού, αλλά προβλέπεται και ένα αυτόματο τέτοιο από το σύστημα. Έτσι γίνονται οι προτάσεις για το τέριασμα ανάδοχο και νέο επιχειρηματία. Τώρα, ε, συμφωνία των στόχων, διάρκεια της επαφής, ε, δραστηριότητες και φυσικά ένα έγγραφο με τις υποχρεώσεις που υπογράφεται σε πρόωρο στάδιο. Το τέταρτο βήμα είναι η παραμονή στην Αλοδαπή. Ε, μια επιτόπου υποστήριξη για τον Ισπανό ε, επιχειρηματία μέσω του γερμανικού ενδιάμεσου οργανισμού. Έτσι μπορούν να καλυφθούν κάποιε δυσκολίε που αντιμετωπίζουν νέε επιχειρηματίε στην αρχή. Και έχουμε και ένα μηχανισμό feedback. Οι επιχειρηματίε ε, απαντούν σε κάποιε ερωτήσει για το πώ μπορεί να βελτιωθεί το πρόγραμμα. Τελική πληρωμή των νέων επιχειρηματιών μετά την επιτυχή διεκπαιρέωση της παραμονής. βέβαια τα έξοδα παραμονής και ταξιδιού ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Ε, κυμαίνονται από 550 με 1.100 ευρώ ανά μήνα για τη διάρκεια της ε, παραμονής. Τώρα για του ανάδοχου επιχειρηματίε, είναι σημαντικό να έχουν αυτού τους ενδιάμεσους οργανισμούς και μάλιστα έχουμε και έναν εκπρόσωπο αυτών των οργανισμών που θα σα μιλήσει στην ακρόαση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε και ένα γραφείο υποστήριξης για το συντονισμό των διοικητικών λεπτομεριών. Επίση θα γίνει μια παρουσίαση και από το γραφείο υποστήριξη. που αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό την αιγύδα των Ευρωπαϊκού, ε, Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων, του Eurocommerce, Eurochamber, συγγνώμη. Και πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέσσερα λοιπόν είναι τα βήματα των ανταλλαγών. Η, ε, η ηλεκτρονική αίτηση, το τέριασμα, η σύναψη της σύμβασης προετοιμασία και η παραμονή στην αλλοδαπή. Τώρα, αναμενόμενα αποτελέσματα και γιατί μπαίνουμε σε όλο αυτόν τον κόπο. Πολλά είναι τα πλέον εκτίματα του προγράμματος Έρασμος για τους νέους επιχειρηματίες. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, ο προϋπολογισμός που έχουμε επιτρέπει ανταλλαγές 500 ε, με 700 το χρόνο επιχειρηματιών. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος και στην πιλωτική φάση είχαμε κάποια προβλήματα, αλλά τώρα έχουμε ρονταριστεί για να επιτύχουμε αυτό το ποσοστό. Επίσης θέλουμε να ενισχύσουμε την δημιουργία νέων επιχειρήσεων και φάνηκε από μια μελέτη και αξιολόγηση ότι μπορούμε να πετύχουμε ένα 20% επιπλέον, επιπλέον δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Επίσης θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα αυτών των επιχειρήσεων. Γιατί οι επιχειρηματίες όταν ξεκινάμε επιχείρηση αισθάνονται πολύ μεγαλύτερη ε, εμπιστοσύνη και σιγουρία εφόσον έχουν συμμετάσχει αυτό το πρόγραμμα. Επίσης, 35% των αναδόχων επιχειρηματιών αυξάνουν την διεθνή τους παρουσία μετά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, άρα είναι και για αυτούς επωφελές το πρόγραμμα. Επίσης, θέλουμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και κατά μέσο όρο νέες επιχειρήσεις δημιουργούν 4,1 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης ε, το χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε είναι προς το συμφέρον όλων να έχουμε νέες ε, επιχειρήσεις. Μειώνεται ε, το περιθώριο αποτυχίας, το ποσοστό αποτυχίας και έχουμε και περισσότερη καινοτομία. Και πάνω από τους μισούς επιχειρηματίες δηλώνουν ότι μετά την παραμονή τους στην Αλοδαπή αυξάνουν κατά πολύ Τη καινοτομία και τις νέες δραστηριότητε. Τώρα, μετά από μια πρώτη πενταετία λειτουργία του προγράμματο μπορούμε να κάνουμε ένα απολογισμό. Πάντως, στην πρώτη αξιολόγηση που έγινε μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργία, φάνηκε ένα υψηλότερο δυναμικό αυτού του προγράμματο. Και το ποσό που απαιτείται από κάθε νέα θέση απασχόληση είναι πολύ ανταγωνιστικό. Κάτω από 10.000 ευρώ για κάθε νέα θέση που δημιουργείται. Οπότε και από αυτή την άποψη το πρόγραμμα είναι πολύ αποτελεσματικό και τα χρήματα του πιάνουν τόπο. Τώρα τα αποτελέσματα εντάχει. Μπορείτε να εξετάσετε δελεχώς τον πίνακα. Έχουμε 7.000 ε, μέχρι στιγμής επιχειρηματίες που έχουν καλυφθεί από το πρόγραμμα. 50% μείωση, ποσοστό μείωσης των επιχειρηματιών που δεν πληρούν τα κριτήρια. Ένα στους 5. Οι υπόλοιποι συμμετέχουν με επιτυχία. Επίσης, αύξηση κατακόρυφη των σχέσεων μετά την καταγραφή. Το πιο ενδιαφέρον είναι οι επιτυχείς σχέσεις και βλέπετε από την καμπύλη πόσες έχουν ευοδοθεί. Έχουμε μια σταθερή αύξηση λοιπόν και έχουμε αυτή τη στιγμή 1.400 σχέσεις που έχουν ολοκληρωθεί. 2.800 ε, επιχειρηματίες δηλαδή γιατί είναι δύο τα μέρη σε αυτή τη σχέση και αυξανόμενος ε, αριθμός, η πρωτοκαλή γραμμή των ε, τρεχουσών σχέσεων που δεν έχουν, των εκκρεμών που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε 280 ε, σχέσεις που πρόκειται να ολοκληρωθούν, δηλαδή 280 νέοι επιχειρηματίες που βρίσκονται στην Ελλαδαπή και συνεργάζονται με έναν ανάδοχο επιχειρηματή. Κάθε εβδομάδα έχουμε 50 με 70 νέες ε, εγγραφές. Οι εγγραφές γίνονται από πολλές χώρες και στοχεύουν σε πολλές χώρες και μάλιστα ο πίνακας φαίνεται άνισος. Βλέπετε το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για το Ηνωμένο Βασίλειο εξαιτία της γλώσσας ε, σε μεγάλο βαθμό. Οι περισσότεροι νέοι επιχειρηματίες θέλουν να πάνε στη Μεγάλη Βρετανία και ανάδοχοι επιχειρηματίε τη Μεγάλη Βρετανία. Ε, ε, ανάδοχοι επιχειρηματίε ενδιαφέρονται για νέου επιχειρηματίε από τη Μεγάλη Βρετανία. Δεύτερη χώρα σε ενδιαφέρον είναι η Γερμανία. Και μετά η συνήθι συχνότητα. Ανάλογα και με το μέγεθο τη χώρα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, υψηλά επίπεδα ενδιαφέροντο και Σουηδία, Βέλγιο, Αυστρία. Ζωηρό ενδιαφέρον λοιπόν από πολλέ χώρε. Οι μικρότερε χώρε δεν έχουν ε, εξοικειωθεί με το σύστημα, γι' αυτό και δεν εκπροσωπούνται δεόντως. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε επίσης μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ της αποτελεσματικότητας των ενδιάμεσων οργανισμών που κάνουν αυτό το τέριασμα των νέων με τους ανάδοχους επιχειρηματίες. Βλέπετε τρεις και στους πιο αποτελεσματικούς θέλουμε ε, όλοι να βελτιώσουν τη λειτουργία τους και καλύπτεται ευρύτατο το φάσμα τομέων. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Ο τομέας των υπηρεσιών ε, υπερεκπροσωπείται σε σχέση και με τις νέες επιχειρήσεις. Κάτι που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί είναι ο μεγαλύτερος τομέας. Επίσης, θέλουμε νέους επιχειρηματίες με επαγγελματική πείρα. Δεν θέλουμε η πλειοψηφία των δικαιούχων να είναι φοιτητέ απλώς. Πάνω από 50% των επιχειρηματιών έχουν τουλάχιστον ένα χρόνο επαγγελματική πείρα. Βέβαια έχουμε και νέους επιχειρηματίες, τελείως και νέους, αλλά 8% των ετούντων έχουν πάνω από δεκαετή πείρα επαγγελματική και αυτή είναι φυσικά ευπρόσδεκτη. Τώρα, ε, βλέπετε για τους ανάδοχους επιχειρηματίες ότι 80% έχουν κάτω από 20 εργαζόμενους. Οπότε ανταποκρίνεται ε, στην αίτησή μας να, δίνεται, να δίνονται ρεαλιστικές πληροφορίες στον νέο επιχειρηματία και τώρα τις πηγές ε, πληροφορίας. Οι ενδιάμεσοι οργανισμοί έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ως πηγή πληροφόρησης γιατί κάνουν και την πρόθεση και το, το, βέβαια το site μας, το σελίδα, αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Τώρα το feedback σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι θετικό από τους νέους επιχειρηματίες. 95% των νέων επιχειρηματιών κρίνουν το πρόγραμμα εξαιρετικά χρήσιμο. Στο δεύτερο πίνακα έχετε το πολύ χρήσιμο και στη δεύτερη γραμμή το χρήσιμο. Θεωρούν πολύ χρήσιμο δηλαδή το πρόγραμμα για να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους. Και βλέπετε ότι πολλοί επιχειρηματίες ε, αμέσως μετά την επιστροφή τους θέλουν να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους. Ήταν ήδη έτοιμοι και θέλουν το συντομότερο δυνατόν να ξεκινήσουν το πολύ μέσα σε ένα χρόνο. Τώρα για τους ανάδοχους επιχειρηματίες έχει παρατηρηθεί και εδώ μεγάλο ποσοστό που είναι εντυπωσιακό γιατί είναι θελοντική η συμμετοχή ε, άνευ αποδοχών αλλά η ικανοποίησή τους είναι μεγάλη κάτι που είναι πολύ θετικό. Τώρα, για τις νέες δραστηριότητες των νέων αναδόχων, των αναδόχων επιχειρηματιών αφορά νέες αγορές, ε, νέες ε, δραστηριότητες, συζήτηση του επιχειρηματικού μοντέλου και ούτως και ούτω καθεξής. Τώρα έχουμε εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των ανταλλαγών. Βλέπετε το 2009 στην αρχή ήταν χαμηλό το ποσοστό των ανταλλαγών, τώρα έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό ρυθμό και με τον προϋπολογισμό μας νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο έπακρο των ανταλλαγών που μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε. Για να τις αυξήσουμε θα χρειαστεί και αύξηση του προϋπολογισμού. Τώρα έχουμε τήσια προκήρυξη για κάθε κύκλο για δημοσιονομικούς λόγους και έλεξε ε, πριν από, δύο, από μία εβδομάδα ο προπολογισμό 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίω, 91 προτάσει έχουν υποβληθεί, 35 εκατομμύρια ε, οι αιτήσει για χρηματοδότηση, 35 εκατομμύρια αιτήσει για χρηματοδότηση. Η μισή φαίνεται ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Αλλά και εξαιτία του προπολογισμού δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες τις αιτήσει. Κάτι που είναι ε, κρίμα δυστυχώς. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε αύξηση του προπολογισμού προκειμένου να ικανοποιήσουμε όλους τους ετούντε. Εν κατακλείδη θα ήθελα να πω ότι ήταν επιτυχές το πρόγραμμα, δύσκολη κάπως η αρχή γιατί είχαμε αρκετές δυσκολίες που έπρεπε να ξεπεράσουμε. Γιατί και το έρασμος είναι σαν επιχειρηματική δραστηριότητα. Υπάρχει ιδέα, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί και να λειτουργήσει. Επίσης, καταπληκτικό το feedback και από τους νέους και από τους ε, αναδόχους επιχειρηματίες. Φαίνεται ότι επηρεάζεται θετικά και ανταγωνιστικότητα και ως προς τη διεθνοποίηση και την καινοτομία η αρχική έκθεση αξιολόγηση ήταν θετική. Έχουμε μια καλή βάση για το μέλλον και επίσης έχουμε και μια άμεση λύση για το πρόβλημα της ενεργείας των νέων, γιατί πραγματικά βοηθούμε τους νέους να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση και να δημιουργήσουν και νέες θέσεις εργασίας. Οι προκλήσεις τώρα ποιες είναι. Καταρχήν έχουμε μεγάλες διαφορές στις επιδόσεις των ενδιάμεσων οργανισμών. Οπότε θα πρέπει να βελτιώσουμε τη δικτύωση για να ανταποκριθούν στα, στις προδιαγραφές ποιότητας. Έχουμε καταρτήσει και ένα εγχειρίδιο ποιότητας και το Σεπτέμβριο ε, θα έχουμε μια πρωτοβουλία για την κατάρτιση ενός κώδικα συμπεριφοράς για το τι αναμένουμε δηλαδή από τους ενδιάμεσους οργανισμούς ώστε να βελτιωθούν και να ανταπεξέλθουν στις υποκρεώσεις τους. Για το θέμα είναι η συνεργασία. Κανένας οργανισμός μόνος του δεν θα μπορέσει να τα καταφέρει. Γι' αυτό θα πρέπει να βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ τους για να καλύψουν και το έδαφος όσοι υστερούν. Επίσης, πρέπει να συγκεντρώσουμε απαιτήσει, ε, μια κρίσιμη μάζα προϋποθέσεων και απαιτήσεων. Φυσικά δεν πρόκειται να ικανοποιήσουμε όλες τις προσδοκίες γιατί υπάρχουν και δημοσιονομικά προβλήματα εξαιτία του περιορισμένου προπολογισμού αλλά και σε ό,τι αφορά του ανθρώπινου πόρου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζεται για να περιορίσει όλο και περισσότερο το προσωπικό τη, κάτι που επηρεάζει και το μέλλον του προγράμματο. Στο μέτρο που θέλουμε να αναπτύξουμε νέε ιδέε και να το επεκτείνουμε. Τώρα, άλλε προκλήσει θέλουμε αυτοί οι ενδιάμεσοι οργανισμοί να καταλάβουν τι απαιτείται από αυτούς, χρειάζεται και δέσμευση και πολλές ε, δεξιότητες και προσόντα. Και φυσικά πολλοί ενδιάμεσοι οργανισμοί θα χρειαστούν απαραίτητη κατάρτιση. Δεν έχουμε εθνικού συντονιστέ δυστυχώ. Αλλά αυτό έχει και πλονεκτήματα και μειονεκτήματα. Θα δούμε αν στο μέλλον ε, αυτό βοηθήσει περισσότερο να βελτιώσουμε τον, το συντονισμό. Υπάρχει μια λεπτή ισορροπία μεταξύ των προσπαθειών για την προώθηση του συστήματος, ε, του προγράμματος και της προσπάθειας ε, ταιριάσματος των επιχειρηματιών. Θα πρέπει να βρούμε το σωστό μείγμα σε όλα αυτά. Τώρα το έρασμος ε, έχει, έχει πια, αποτελεί πια ένα απόσπαστο τμήμα του κόσμου. Υπάρχει ε, για την πρώτη πενταετία ένα σχέδιο αξιολόγηση ήδη και υπάρχει μια πρόταση για διεύρυνση του προπολογισμού. Θα κάνω μια εξωτερήκευση του προγράμματος προς την Οργανισμό για την Καινοτομία και ε, την επιχειρηματικότητα στις αρχές του επόμενου έτους και επίσης έχουμε ε, και τα γραφεία στήριξης για την καθημερινή διαχείριση του προγράμματος και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε αύξηση των συνεργειών χάρη σε αυτή τη διαδικασία εξωτερήκευσης που κάνουμε αλλά δεν πρόκειται να γίνει μια συγχώνευση με το δίκτυο επιχειρηματιών. Επίσης, θέλουμε να δημιουργήσουμε και μία ομάδα εργασίας για να δούμε τι βελτιώσεις ε, μπορούν να γίνουν, να βρούμε τα προβλήματα, τις θενοπούς, ώστε να μπορέσουμε να επιταχύνουμε την αποτελεσματικότητα του προγράμματος και να φτάσουμε σε 10.000 ε, ανταλλαγές το χρόνο μέχρι το 2020, που δεν είναι τόσο μακριά όσο ακούγεται, όσο φαίνεται, αυτή τη στιγμή έχουμε 2.000 ανταλλαγέ το χρόνο εξαιτία του περιορισμένου προπολογισμού, αλλά θα πρέπει να βελτιώσουμε το έργο, τα, τα εργαλεία που έχουμε. Όλα αυτά θα τα εξετάσουμε εντελεχώ και ελπίζω η σχετική έκθεση αξιολόγηση να δημοσιευθεί μέχρι τα μέσα του 2014. Να μπορέσουμε να κάνουμε μια γενική επισκόπηση του προγράμματο των επιμέρου στοιχείων του και νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε χαρίς για το ότι ξεκίνησε αυτή η συνεργασία και ευχαριστούμε θερμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη που μας έδωσε στο πρόγραμμα αυτό που εξυπηρετεί και τους νέους επιχειρηματίες αλλά και βελτιώνει την απασχόληση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ και είμαι στη διάθεση της ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Μετά τους ομιλητές θα τεθούν τα ερωτήματα. Ο επόμενος ομιλητής, η κυρία Μικαέλα Παντίνη υπεύθυνη της RCD αρχιτεκτούρα στην περιοχή της Ματέρα της Ιταλίας και ήταν πολλές φορές ε, φορές υποδοχής νέων επιχειρηματιών βάσει του προγράμματος Εράσμους για επιχειρηματίες. Θα σας ακούσουμε για ό,τι έχει να μας πείτε. Uh, good morning. Thank you very much for the invitation. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε την εδώ στην πόλη της Ματέρα, στην Ιταλία. Διστάζαμε στο ξεκίνημα να μπούμε στη διαδικασία του Erasmus ε, Entrepreneurship, γιατί δεν είδαμε ένα άμεσο δεν είχαμε δει ένα άμεσο κέρδος για την επιχείρηση. Ξεκινήσαμε πριν από 1,5 χρόνο με τον πρώτο επιχειρηματία που ήρθε στη Ματέρα. Η Ματέρα είναι μια μικρή, μικρή πόλη στην Νότια Ιταλία με πολλή ανεργία, περίπου 40% ανεργία των νέων. Έχει 55.000 κατοίκους, έχει ένα πολύ όμορφο, μια πολύ όμορφη περιοχή που είναι που έχει κηρυχθεί η πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας από την UNESCO. Είχαμε ένα προπολογισμό για τους νέους επιχειρηματίες, γύρω στα 800 ευρώ έπαιρναν τον χρόνο. Ε, βρήκανε στέγη, ένα δωμάτιο στην πόλη θα είχε πάνω από, δεν κόστιζε πάνω από 200 ευρώ, οπότε είχαν ήταν πλήρη η κάλυψη, δεν χρειαζόταν να ενταχθεί σε, άλλου σε άλλους πόρους. Έχει πανεπιστήμιο η πόλη, έχει ένα νέο, ένα νέο κάμπους για τους πανεπιστημιακούς φοιτητές. ενώ τώρα είναι υποψήφια για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα για το 2019. Τώρα, σε μια μικρή πόλη οι επιχειρηματίες και οι τρεις εμπειρίες που είχαμε δηλαδή είχαν τη δυνατότητα να ενταχθούν πλήρως στην κοινωνική ζωή της πόλης. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Μια μικρή πόλη σημαίνει ότι ζούσαν και δούλευαν μαζί μας, περπατούσαν πέντε λεπτά, λεπτά από το σπίτι στη δουλειά, μπορούσαν να γίνουν κομμάτι της πόλης και να ζήσουν την εμπειρία τους. Τρεις ξένοι ήρθαν και έμαθαν τη ματέρα και την Ιταλία πολύ καλά. Οι βασικές ε, δραστηριότητε είναι ε, μικρά ταξίδια. Είμαστε μικρή επιχείρηση, δουλεύουμε με προγράμματα, marketing και δικτύωση έργων με outsourcing σε καμιά δεκαριά, 20 άτομα. Στο γραφείο ήταν τρία άτομα. Δουλεύαμε με το Viaggio Architecture που είναι μια online εταιρεία επισκέψεων ε, για αρχιτέκτονες στη Νότια Ιταλία. Το Sassy Web που είναι μια επιχείρηση ε, που δουλεύει στην Ματέρα. Το Can't Forget Italy, ένα άλλο project που έχει οπτικό περιεχόμενο για την προώθηση της Ιταλίας ε, και το Expo του Μιλάνου 2015. Δύο από τους ε, φοιτητές του Εράσμους είχαν, εμπλαχθεί, είχαν συμμετάσχει στα δύο τελευταία έργα. Οι υποψήφοι ήταν από την Ολλανδία, την Ουγγαρία και τη Σουηδία. Ο πρώτος υποψήφιος ήταν ο Κάσπερ από την Ολλανδία. Δούλεψε έξι μήνες στα γραφεία μας και ήθελε να ξεκινήσει μια επιχείρηση που θα έλεγε οπτικές ιστορίες οπτικές ταξιδιωτικές ιστορίες με αμοιβή. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε μαζί. Είχε έρθει με ένα μικρό, με μια μικρή Sony βίντεο κάμερα. Ξεκινήσαμε να γράφουμε, να φτιάχνουμε τις, τις ταξιδιωτικές διηγήσεις μας μαζί. Τον πρώτο χρόνο μετά το Εράσμους μπορέσαμε να του αναθέσουμε συμβόλαια αξίας 20.000 ευρώ περίπου, είτε άμεσα εμείς, είτε μέσω επιχειρήσεων που μας έδιναν τις, ε, που μας ανέφεραν προγράμματα. Δηλαδή έκανε τη δουλειά που ήθελε να κάνει, έλεγε ταξιδιωτικές ιστορίες. Προφανώς μπόρεσε να αναβαθμίσει τον εξοπλισμό του, έγινε επιχειρηματίες. Ε, μάλιστα ζει τώρα στη Ματέρα, ήρθε εδώ μετά το έργο και δουλεύει μια χαρά. Αυτό είναι success story. Δε, ο δεύτερος υποψήφιος, υποψήφια ήταν μια Ουγγαρέζα. Ένα μήνα έμεινε μαζί μας μόνο δυστυχώς. Και αν θέλω να κάνω μια επικοδομητική κριτική, ο ένας μήνας δεν αρκεί. Δεν αρκεί για να ξεκινήσει κάποιος να δουλεύει για κάτι μακροπρόθεσμο, τουλάχιστον σε δικό μας επίπεδο. Η συνάδελφη ήταν πολύ καλή κοπέλα, δούλευε για ένα project ψηφιακού ημερολογίου και ήταν ε, διευθύ, ε, ε, σκηνοθέτης ενός ε, φιλμ που είχαμε ετοιμάσει για την περιοχή του Μπαζιλικάτα. Η Ιζαμπέλ Πάλο έφυγε πριν από λίγο. Η Ιζαμπέλ δούλεψε για τρεις μήνες. Είναι μουσιογράφος από την Σουηδία. Δεν ήξερε τι ήθελε να κάνει. μας ε, βοήθησε να καταλάβουμε το μηχανισμό του πώς φτιάχνεις και τοποθετείς μία ιστοσελίδα. Η Ιζαμπέλ βοήθησε να δημιουργήσει, ανέλαβε το Milan Expo του στα χέρια της και έγραψε πολύ όμορφα κείμενα, είχε, κάνει καλές μετα... είχε ε, αποκτήσει καλές μεταφράσεις και σιγά σιγά της εξηγούσαμε πώς φτιάχνεται μια ιστοσελίδα, πώς γράφεις τις λέξεις κλειδιά και το περιεχόμενο για να έχεις ένα αποτελεσματικό, μια αποτελεσματική ιστοσελίδα. Το έργο πήγε πολύ καλά, έχει μεταφραστεί στα κινέζικα όπως βλέπετε και έκανε συντονισμό των μεταφράσεων, τα πάντα. Κάτι άλλο που είδα στην περίπτωση της Ιζαμπέλ ότι προφανώ το Μιλάν Expo του μιλάει για το Μιλάνο. Έχοντα δουλέψει τρει μήνες και έχοντα γράψει τρει μήνες για το Μιλάνο, σκέφτηκα ότι θα τον ωραίο να τη στείλω στο Μιλάνο. Και οργανώσαμε ένα ταξίδι να πάει να δει τι είναι το Μιλάνο. Δεν υπήρχε ασφάλιση ασφαλιστική κάλυψη για κάτι τέτοιο. Και ξέρετε, η δική μας ε, κατηγορία επιχειρήσεων είναι κινητική. Πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί. Θα βοηθούσε λοιπόν πάρα πολύ να μπορέσουμε να έχουμε ασφάλιση για τα άτομα αυτά, όχι μόνο στο γραφείο, αλλά και για κάποια κομμάτια των ταξιδιών τους. Τι μάθαμε τώρα. Σίγουρα είναι μια θετική εμπειρία για μας. Δουλεύοντας με ταξιδιωτικά project, βλέπουμε ότι πολλοί άνθρωποι που έρχονται και ξεκινούν να δουλεύουν σε δικά μας έργα, βλέπουν πράγματα που εμείς δεν βλέπουμε. Εμείς δουλεύουμε με ιδέες και προγράμματα για ιστοσελίδες 6-7 μήνες και συχνά δεν βλέπουμε προβλήματα. Δεν βλέπουμε λάθη. Κάποιος που έχει τα παίξω, ως χρήστης ή ως ε, ξένος από το πρόγραμμα μας βοηθά να βελτιώσουμε, να σκεφτούμε καλύτερα και να βελτιώσουμε ένα κείμενο. Ήταν πολύ σημαντικό. Η διάδραση με, το, με τους νέους επιχειρηματίες ήταν πολύ σημαντική στην πόλη. Η δυνατότητα που είχαν να μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους σε άλλους και μέσα στο γραφείο και έξω από το γραφείο ήταν πολύ σημαντική. Εμείς δουλεύουμε σε μια πολύ συγκεκριμένη σε ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς που πάει καλά στην Ιταλία αλλά υπάρχουν κενά στην, ε, στον κλάδο των ταξιδιωτικών ε, υπηρεσιών όπου θα μπορούσαμε, θα να εκμεταλλευτούμε καλύτερα και να κερδίσουμε όπως κάποιοι νέοι επιχειρηματίες. Μια win-win κατάσταση λοιπόν, κερδίζουν και οι δύο. Ο κύριος Βάινμπεργκερ είπε ότι δεν έχουμε αμοιβή. Οι επιχειρήσεις δεν ε, αμείβονται. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ ωστόσο έμαθα πάρα πολλά πράγματα και με βάση το πρόγραμμα Εράσμους και την εμπειρία ε, μπορέσαμε να δημιουργήσουμε νέες ε, εγκαταστάσεις που θα ξεκινήσουν τον άλλο μήνα με καλύτερα γραφεία όπου θα έχουμε όχι μόνο φοιτητές Εράσμους αλλά φοιτητές σε ανταλλαγή από ολόκληρο τον κόσμο. Ε, στην ίδια περιοχή έχουμε 20 θέσεις εργασίας αλλά και ένα διαμέρισμα όπου μένουν οι, όσοι εμπλέκονται σε ε, ένα πρόγραμμα ανταλλαγή. Άρα μπορούμε να στεγάσουμε με μηδέν κόστος κάποιον ε, νέο επιχειρηματία ή κάποιον φοιτητή που δεν χρηματοδοτείται από κάτι άλλο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι η εικόνα που έχουν άλλοι ότι μπορούν να φέρουν, αυτό που μπορούν να φέρουν οι διεθνεί διάστασει που μπορούν να φέρουν στο επιχείρημα είναι πολύ ζωτική. Δεν ξέρω αν θέλετε, αν σα ενοχλεί που κλείνω ε, με μια πρόταση τη γουίνι, τη Αρκούδα. Δεν, μπορεί να μην, ε, μπορείς να μείνεις ε, στη γωνιά στο δάσος περιμένοντας οι άλλοι να έρθουν σε σένα. Πρέπει να πας εσύ σε αυτούς μερικές φορές. Ευχαριστώ και ευχαριστώ που επιτρέψατε να συνεχίσουμε και τις επόμενες, ε, την επόμενη περίοδο με νέους επιχειρηματίες. Σας ευχαριστώ και νομίζω ότι τώρα θα ζητήσουμε από τους τεχνικούς να προβάλλουν την ταινία. Technik wird in einigen Minuten das gewährleisten. Σε λίγα λεπτά θα το καταφέρουμε να, το, να προβάλλουμε την ταινία.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 Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την, ε, το Euronews που μας ε, δείχνει έτσι διάφορα επίκαιρα θέματα. Και έχουμε εδώ πέρα και τον τηλεοπτικό μας αστέρα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως ε, που έχουμε μαζί μας τον κύριο Λιμπίδας Μπούτκους, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το Βελομπλικ στην Κλαπέντα. παρευρέθηκε στην ε, Αυστρία για κάποιους μήνες ως νέος επιχειρηματίας. Καλώς ορίσατε λοιπόν, να σας ακούσουμε. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Ρίμιτα Ζεμπούτκους. Το 2009 συμμετείχα στο πρόγραμμα Εράσμους για νέους επιχειρηματίες και στο κράτος της Αυστρίας ε, μετέβησα. Έμαθα για το πρόγραμμα αυτό κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας επιχειρηματικότητας. Και κατάλαβα ότι για να βρει κανείς ε, επαφές θα πρέπει να είναι αποφασισμένος. Και φυσικά πολλά εξαρτώνται και από τον παράγοντα της τύχης. Συμμετείχα σε σεμινάρια, σε παρουσιάσεις για επιχειρήσεις. Ήταν δύσκολο να κάνω επαφές γιατί Ξέρετε, εγώ μιλούσα μόνο γερμανικά ως ξένη γλώσσα, άρα μόνο στην Αυστρία και την ε, Γερμανία εξέτασα ως ε, ενδεχόμενο. Ξεκίνησα λοιπόν ψάχνοντας μια οργάνωση η οποία θα μπορούσε να με βοηθήσει. Έστειλα email, επιστολές Επίσης προσέγγισα διάφορες ε, ενδιάμεσες ε, οργανώσεις και στην Αυστρία και στη Γερμανία και κατάφερα να θέσω τις πρώτες επαφές ουσιαστικά με μια εταιρεία στο Κράτς. Ήταν περίπλοκη ωστόσο η κατάσταση γιατί έστελνα ηλεκτρονικές επιστολές οι οποίες κατέληγαν στο spam, στο κάδο απορριμμάτων της ε, εταιρείας και πολύ απλά δεν τα έβλεπε κανείς τα γράμματα μου. Ουσιαστικά κατά σύμπτωση Τελικά έφτασε μία επιστολή μου ηλεκτρονική και τελικά δημιουργήθηκε μία επαφή. Μέσω της επαφής αυτής κατάφερα να προσεγγίσω τις ενδιάμεσες οργανώσεις, την ενδιάμεση οργάνωση στην Αυστρία. Στην αρχή να σας πω, ήταν όλοι πάρα πολύ φιλικοί μαζί μου. Θεωρώ ότι αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι είχαμε την ίδια ηλικία, ότι ήμασταν ευγενικοί ο ένα με τον άλλον και νομίζω ότι στο μέλλον αυτό θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα. Είναι απαραίτητο να επενθυμίζουμε στις εταιρείες που φιλοξενούν ότι πρόκειται για ένα άτομο το οποίο θα πρέπει να το βοηθούν. Και αυτός ο νέος επιχειρηματίας θα πρέπει επίσης να κατανοεί πότε μπορεί να δώσει ο ίδιος κάποια σύσταση, κάποια συμβουλή και πότε θα πρέπει να σιωπήσει και να απορροφήσει αυτά που βλέπει. Το πρόγραμμα αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, θεωρώ, γιατί δίνει μεγάλες δυνατότητες να εξοικειωθεί κανείς με πάροχους ε, υπηρεσιών. Το 2001 είδα στο Αμβούργο, στη Γερμανία, έναν κούριερ με, ποδηλά, με ποδήλατο. Και πραγματικά ε, βρήκα συναρπαστική την ιδέα. Γι' αυτό λοιπόν επανήλθε αυτό το 2009. Η δυνατότητα γρήγορης χρηματοδότησης αποτέλεσε και έναν από τους λόγους για τους οποίους αποφάσισα να συμμετέχω στο πρόγραμμα αυτό. Ιδάλλως θα ήμουν ακόμα υπάλληλο. Νομίζω ότι αυτή η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι πάρα πολύ σημαντική για νέους επιχειρηματίες. Επίσης, ε, η εταιρεία υποδοχής, να σας πω ότι και αυτή επωφελείται από το πρόγραμμα, γιατί ουσιαστικά εξετάζει την επιχείρηση από ένα νέο πρίσμα, μέσα από ένα νέο πρίσμα. Και ο νέος επιχειρηματίας ασφαλώς και μπορεί να προσφέρει και αυτός την εμπειρία του τις συμβουλές του. Είναι επίση δυνατή η ανταλλαγή επιχειρηματικών ιδεών. Έχω δει τρεις επαφές, ξέρετε, με την εταιρεία υποδοχή για ένα νέο επιχειρηματία. Επίσης είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορούν να εξετάσουν νέοι σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο εκ των έσω, χωρίς να χρειαστεί να επαναφεύρουν τον τροχό. Έτσι εμπνέεται κανείς μαθαίνει τη δουλειά στην πράξη και έτσι είναι πιο εύκολη ενδεχομένως η σύσταση μια δική του επιχείρηση μετά. Επίσης αποκτά τεχνολογία αχμής αν θέλετε. Στην δική μου χώρα εισήγαμε ουσιαστικά μια νέα υπηρεσία σε ό,τι αφορά τη μεταφορά πακέτων με ποδήλατο. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η υπηρεσία courier ήταν πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμη, πάρα πολύ πολλά υποσχόμενη για το μέλλον. Θέλουμε να επεκταθούμε τώρα σε άλλες πόλεις. Θέλουμε να απασχολήσουμε φοιτητέ που μπορούν να δουλέψουν κάποιες ώρες την ημέρα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να προωθηθεί το πρόγραμμα αυτό το δίχως άλλο και σε μεγαλύτερη κλίμακα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και θα έπρεπε να μιλήσουμε σε σχολεία, ε, πανεπιστήμια, σχολές, ε, οργανώσεις. Θα πρέπει να δημιουργηθούν σύνδεσμοι και επαφές μεταξύ των ε, τοπικών εταιριών και των συντονιστών. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο κύριος Ρουμπίχη, ο Πρόεδρος. Ήταν πάρα πολύ καλό και χρήσιμο αυτό το πρακτικό παράδειγμα. Αυτό το πρακτικό παράδειγμα που έχει στεφθεί με επιτυχία. Τώρα περνάμε στο επόμενο, σύντημα, στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Το δίκτυο υποστηρίξης. Καλώς ορίζω τον κύριο Αρνάλντο Απροτσίνη, ο οποίος είναι Γενικός ε, Γραμματέας του Eurosamps των Ευρωπαϊκών ε, Επιμελητηρίων και θα του δώσω το λόγο παρά αυτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, το Eurochambers, τα επιμελητήρια, οργανώνουν μια σειρά προγραμμάτων από την Ευρώπη με πολλέ δραστηριότητε. Ένα όμως από τα προγράμματα για τα οποία είμαστε περήφανοι είναι το Εράσμος για νέους επιχειρηματίες. Ανάλογα με την προοπτική που θέλετε να το δείτε από την οπτική της απασχόλησης, της νέας επιχειρηματικότητας, της νέας δημιουργίας θέσεων επιχειρήσεων, της συμβολής στον πλούτο μιας χώρας, το Εράσμος δίνει ούτως ή άλλως απάντηση. Και γι' αυτό από την αρχή του προγράμματος βοηθήσαμε την ανάπτυξη του προγράμματος. Από την επινόησή του μπορεί να έχουμε τα, τα φώτα κάτω. Από την δημιουργία του προγράμματος το 2007 σαν αποτέλεσμα μεγάλου λόμπι και συζητήσεων που είχαμε ως ε, ε, επιμελητήρια με, το, την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά τη δημιουργία του Εράσμους για τους ε, νέους επιχειρηματίες ήμασταν πάντα υπεύθυνοι και ως Ευρωπαϊκό Συντονιστικό Γραφείο και ως ενδιάμεση. Θα δείτε ότι μοιράσαμε την ιστορία του προγράμματος σε τέσσερις σε τέσσερα στάδια. Και αυτό είναι χρήσιμο γιατί μπορούμε να δούμε τι βελτιώσεις μπορούμε να περιέχουμε σε κάθε διαμόρφωση, μελλοντική διαμόρφωση του προγράμματος. Το startup, το ξεκίνημα, η πρώτη περίοδος του προγράμματος. Η κατασκευή του προγράμματος στην ουσία που ήταν το παραδοσιακό Στηρίζοντα το παραδοσιακό εράσμο των φοιτητών που δίνει αμέσως και ο τίτλος δηλαδή δίνει αμέσως την εικόνα της κινητικότητας. Ο πρώτος στόχος ήταν λοιπόν το ξεκίνημα δραστηριοτήτων. Και στηριζόταν ότι για να είσαι καλός επιχειρηματίας πρέπει να έχεις μια κάποια εμπειρία. Με προπόνηση σε κατά κάποιο τρόπο για να γίνεις καλός επιχειρηματίας. Ο στόχος λοιπόν, η βασική κατευθυντήρια γραμμή αυτής ήταν αυτός ο στόχος. Κατόπιν, η δεύτερη φάση, το δεύτερο στάδιο, ήταν η ποσότητα. Το να πάρουμε αυτούς που είναι και ικανοί και ικανοί να δημιουργήσουν θέσεις και ικανοί να εκπαιδεύσουν αυτούς. Αυτό περιέχει και την δημιουργία ενός δικτύου ενδιάμεσων οργανώσεων ανά την Ευρώπη που θα μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά αυτή. με μικρή κατανόηση της τοπικής κατάστασης στις χώρες και περιοχές μας. Γι' αυτό το δίκτυο των ενδιάμεσων ε, οργανώσεων είναι κρίσιμο στοιχείο του προγράμματος. Χωρίς την υποστήριξή τους, το Εράσμους για νέους επιχειρηματίες δεν θα είναι τόσο, τόσο επιτυχημένο. Τρίτη φάση, που είναι αυτό που μπορούμε να πούμε σήμερα, σχετίζεται με την ποιότητα, βελτιώνοντας την κατάσταση, τον αριθμό αυτών που εμπλέκονται και ταυτόχρονα την ποιότητα, βελτιώνοντας την ποιότητα από διάφορες οπτικές. Υπάρχει η ποιότητα του δικτύου, ακούμε ότι η ποιότητα των ενδιάμεσων δομών δεν είναι η ίδια ανά την Ευρώπη, Βελτιώνουμε λοιπόν την ποιότητα των διαδικασιών και την ποιότητα των υποψηφίων και της φιλοξενίας, διότι μπορεί να έχεις μια ανταλλαγή μικρής αξίας που, ή που άλλες ανταλλαγές που έχουν μεγάλη ουσιαστική αξία. Μετά πρέπει να δούμε τις επόμενες εξελίξεις. Κατά την άποψή μας, επόμενη διαφάνεια παρακαλώ, κατά την άποψή μας υπάρχουν κάποια κρίσιμα στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Πρώτον, την αξιολόγηση αυτή καθεαυτή του προγράμματος. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο της Επιτροπής κ. Μπέγκερ, να μιλάει γι' αυτό επί μακρόν. Όντως υπάρχει μια εγενής αξία στο πρόγραμμα η αξιολόγηση λοιπόν όσων μετέχουν στο πρόγραμμα είναι πολύ σημαντική. Μετά έχουμε να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το πρόγραμμα και να πετύχουμε την κρίσιμη μάζα που σήμερα λείπει. Η κρίσιμη μάζα μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους. Είτε με αύξηση του προπολογισμού, είτε με αύξηση της αποτελεσματικότητας. Τα δύο αυτά στοιχεία δεν πηγαίνουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις το ένα με το άλλο. Μπορεί να τα πετύχουμε μαζί. Η αύξηση του προπολογισμού σίγουρα ένα σημαντικό στοιχείο έχει ήδη επιτευχθεί με τη συμπερίληψη του Εράσμους για νέους επιχειρηματίες στο, στον προπολογισμό κόσμο για την επόμενη χρηματοοικονομική περίοδο. Ο προπολογισμό αυτός ωστόσο σύμφωνα με την τωρινή κατανομή των δαπανών και τη σημερινή κατάσταση δεν θα επιτρέψει πάνω από 1500 ανταλλαγές το χρόνο. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά για να φτάσουμε μια κρίσιμη μάζα που η ίδια η Επιτροπή θεώρησε ως σημαντική. Για να έχουμε 10.000 ανταλλαγές το χρόνο δεν φτάνουν τα λεφτά. Πρέπει λοιπόν να βρούμε δημιουργικούς τρόπους για να ζευγαρώσουμε τον προϋπολογισμό αυτό με άλλα κονδύλια. Επίσης θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και στην, στη διάσταση κόστους. Ο υπολογισμός ε, χοντρικά του κόστους μίας ανταλλαγής σήμερα ανέρχεται στα 8 με 10 χιλιάρικα. Αυτά είναι πολλά. Η αύξηση του αριθμού των ανταλλαγών θα βοηθήσει να μειώσουμε το κόστος αναανταλλαγή. Διότι από τις 8 με 10.000 ευρώ τα 50% περίπου είναι δράσεις προώθησης, οργάνωση και διοικητικό κόστος. Το κόστος αυτό δεν θα αυξηθεί αν αυξήσουμε τον αριθμό των ανταλλαγών. Ενώ το άλλο 50% που είναι κονδύλια για νέους επιχειρηματίες θα αυξηθούν ποσοτικοποιημένα. Αυτό θα οδηγήσει σε δραματική αύξηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ο κίνδυνος ότι θα οδηγήσει σε, καλύτερη, σε καλύτερα αποτελέσματα. Κάτι, μια άλλη διάσταση σημαντική όταν πάμε σε ένα νέο επιχειρηματία, το χειρότερο μπορούμε να του πούμε, η χειρότερη εντύπωση που μπορούμε να του δώσουμε είναι ότι για να γίνει επιχειρηματίας πρέπει να μπει σε μια περίπλοκη γραφειοκρατική διαδικασία που δεν τελειώσει ποτέ. Και αν δίνουμε τέτοια εντύπωση στους ε, νέους επιχειρηματίες είναι λάθος. Πρέπει λοιπόν να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες. Με βάση όλους όσοι ζουν στην Ευρώπη η μείωση του διοικητικού βάρους είναι στόχος. Άρα και στη διαχείριση των προγραμμάτων πιστεύω ότι πρέπει να αυξήσουμε την, το να, να μειώσουμε το διοικητικό κόστος που δίνει κόστος που δεν δικαιολογείται για τη λειτουργία του προγράμματος. Δύο προτάσεις για το μέλλον. Εμείς θα, θα μετάσχουμε βέβαια στην αξιολόγηση του προγράμματος στα πλαίσια της ε, επαιτίου του, αλλά θέλω να σας πω κάποιες ιδέες. Πρώτον, παρότι μας είπαν ήδη ότι δεν είναι δυνατή με τα ήδη ε, με τις ήδη λειτουργούσες δραστηριότητες ε, επιτόπου θα έπρεπε να μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση με άλλα δίκτυα όπως το Europe for Entrepreneurship. Είναι ένα δίκτυο που υπάρχει, έχει επαφή με τις, με επιχειρήσεις και δίνει αποτελέσματα. Ήδη έχω, επίσης επι, επαφές έχουν και τα μέλη της των οργανώσεών μας. Το να στηριζόμαστε αποκλειστικά στο ένα δίκτυο δεν αποδίδει. Πρέπει να αυξήσουν τα αριθμό μέσα στο πλαίσιο των υφιστάμενων ενδιάμεσων δομών. Και αυτό σχετίζεται με τη γεωγραφική κάλυψη. Άνηση αυτή τη στιγμή. υπάρχουν πολλές ενδιάμεσες οργανώσεις σε κάποιες χώρες, πολύ λίγες σε άλλες. Η γεωγραφική κάλυψη του δικτύου λοιπόν μπορεί να βελτιωθεί. Τρίτον, υπάρχει ένα στοιχείο με το όνομα του προγράμματος που είναι παραπλανητικό μερικές φορές γιατί μιλάει για νέους επιχειρηματίες και άρα κάποιος μπορεί να νομίσει ότι αυτό είναι ένα πρόγραμμα για 25 άριδες. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η αλλαγή λοιπόν της εικόνας του προγράμματος με ένα νέο τίτλο «Εράσμους για επιχειρηματίες» όπως έχουμε «Εράσμους για φοιτητές». Αυτό θα συμβάλλει και στην αλλαγή της εικόνας του προγράμματος που ξεκινά να είναι ευρύτερα γνωστό τώρα. Και αυτό είναι ο λόγος για το οποίο τα στοιχεία των ανταλλαγών δείχνουν τεράστια αύξηση τους τελευταίους μήνες. Το Εράσμους των φοιτητών 30 χρόνια τρέχει. Τώρα έχουν όνομα στην αγορά. Το Εράσμους για τους νέους επιχειρηματίες δεν έχει αυτό το όνομα ακόμα. Αλλά αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Μια τελευταία παρατήρηση. Ας γίνουμε και πιο δημιουργικοί, συνδυάζοντας νέες εξελίξεις για το εράσμος για νέους επιχειρηματίε. Ξέρουμε ότι ένας από τους βασικούς στόχους των κρατών μελών σήμερα είναι να βρουν νέους τρόπους για να αντιμετωπίσουν, να μειώσουν την ανεργία των νέων, που αυξάνεται με τόσο δραματικό τρόπο σε πολλά κράτη-μέλη η ενεργεία των νέων μπορεί να ειδωθεί από πολλές οπτικές γωνίες. Μία ωστόσο είναι να δώσουμε στον κόσμο την ευκαιρία να δημιουργήσουν τις δικές τους δουλειές. Δεν έχουμε, δεν πρέπει να στοχεύουμε μόνο στην απασχόληση όπως με την παραδοσιακή έννοια, αλλά και σε νέες επιχειρήσεις για να μειώσουμε το ποσοστό ενεργείας αλλού. Αυτό αναφέρθηκε ήδη. Αν όμω το συγκεκριμένο θέμα σημαίνει ότι για παράδειγμα υπήρξαν πολλά κονδύλια που δόθηκαν 6 δις και σε δραστηριότητε που θα πρέπει να αναπτυχθούν σε κράτη-μέλη ή υπό την ευθύνη των κρατών μελών για να μειώσουν την ενεργεία των νέων. Εμείς ήδη συζητούμε άτυπα με ορισμένα κράτη-μέλη για να επαναλάβουμε ένα πρόγραμμα για νέους επιχειρηματίες, χρησιμοποιώντας, χρησιμοποιώντας τα κονδύλια αυτά για να προσθέσουμε δράσεις. Οπότε, δεν θα στηριχτούμε μόνο στις ε, τα κονδύλια του κόσμου που είναι λίγα και παρά τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου δεν πιστεύουν ότι θα αυξηθούν δραματικά στην επόμενη χρηματοοικονομική περίοδο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πόρους που υπάρχουν σε κράτη-μέλη για δύσκολους σκοπούς και δύσκολους στόχους για να αυξήσουμε την ικανότητα του προγράμματος. είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να αλλάξει την άποψη των Ευρωπαίων πολιτών για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπρουτσίνη και τώρα περνάμε στον επόμενο μιλητή, κυρία Αναμαρία Μικέλα, η οποία είναι project manager από τη Φιλανδία, από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων ε, Επιστημών, από το CNOK. Αν υπομονούμε να ακούσουμε τι έχει να μα πείτε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτά, κυρίες και κύριοι. Αισθάνομαι πάση χαρίς για την παρουσία μου εδώ, γιατί εκπροσωπώ όχι μόνο το Σενιόκι, το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Φιλανδίας, αλλά και τους ενδιάμεσους οργανισμούς ε, σε αυτό το πρόγραμμα για τους νέους επιχειρηματίες. Εγώ κατάγομαι από την περιοχή της ε, Νότιας Οστροβόρνιας, της Φιλανδίας. Και είμαστε γνωστοί ε, για την επιχειρηματικότητα. Είμαστε γνωστοί για την επιχειρηματικότητά μας, γιατί μας αρέσει να ανοίγουμε δικές μας επιχειρήσεις. Επικεντρωνόμαστε λοιπόν στο θέμα της επιχειρηματικότητας, γι' αυτό και το πρόγραμμα Έρασμος ε, εντάσσεται πλήρως στους περιφερειακούς μας στόχους που επικεντρώνονται κυρίως στην συνδρομή προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε 17 με 18.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στην περιφέρειά μας. 98% από αυτές είναι πραγματικά πολύ μικρές ε, ή μικρές επιχειρήσεις. Είμαστε η κορυφαία οργάνωση στη με μέλη από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία και την Ιταλία. Και για τον έκτο κύκλο του Έρασμος, για τους νέους επιχειρηματίες, έχουμε διευρύνει τις ε, εταιρικέ μας σχέσεις ε, και καλύπτουμε και τη Σουηδία και την Πορτογαλία στα προγράμματά μας. Ξεκινήσαμε το σχέδιο αυτό, το πρόγραμμα αυτό, ως ε, φιλανδικός ενδιάμεσος οργανισμός, και όπως ακούσαμε και προηγουμένως, είναι αδύνατον να διαχειριστεί κανείς ένα τέτοιο μεγαλεπίβολο πρόγραμμα χωρίς εταίρους σε άλλες περιεφέρειε της Ευρώπης. Γι' αυτό και επεκτείναμε τις εταιρικέ μας σχέσεις προς άλλες χώρες. Και έτσι ξεκινήσαμε. Και αναπτυχθήκαμε. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τους εταίρους μας και τη συνεργασία που έχουμε και με άλλες ενδιάμεσους οργανισμούς. Το πρόγραμμά μας επικεντρώνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Γιατί? Επειδή θεωρούμε ότι στον τουρισμό οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να βελτιώσουν τις ε, πρακτικές τους ε, στο management και χρειάζονται και μια πιο διεθνή προοπτική στις ε, δραστηριότητές τους. Χρειάζονται τις απόψεις και τις αγνώμες και άλλων χωρών σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη προϊόντων και την διάθεση του εμπορία. Επίσης, ε, στηρίζουμε και τις περιφερειακές στρατηγικές για την ανάπτυξη του τουρισμού. Ξεκινώ λοιπόν με μια πολύ αισιόδοξη νότα. Το πρόγραμμα είναι εξαιρετικό με συγκεκριμένους στόχους. Μάλιστα συμμετείχα σε πολλά προγράμματα, αλλά το Erasmus είναι ένα πρόγραμμα που έχει άμεσα αυτά αποτελέσματα για τους επιχειρηματίες. Δεν χρειάζεται να περιμένουν χρόνια ολόκληρα για να δουν αποτελέσματα, αλλά τα βλέπουν αμέσως από τις ανταλλαγές που διευκολύνει το Erasmus. Ε, έχουμε λοιπόν περιπτώσεις επιχειρηματιών ε, που επειδή δεν μπορούν να επαναλάβουν, θέλουν τόσο πολύ να επαναλάβουν την εμπειρία που από ανάδοχοι επιχειρηματίες ε, γίνονται νέοι προκειμένου να επωφεληθούν δεύτερη φορά. Οπότε ο ανάδοχος από τη στιγμή που αφιερώνει μία ώρα στο νέο επιχειρηματία ουσιαστικά λαμβάνει δύο ώρες ε, σε αντάλλαγμα. Δηλαδή το όφελος είναι μεγάλο και για τον ανάδοχο επιχειρηματία, για την επιχείρησή του. Για να αναφερθώ σε επιτυχείς εμπειρίες ε, του προγράμματος, ε, προέρχεται από άλλο ενδιάμεσο οργανισμό της Φιλανδίας, όπου ο νέος επιχειρηματίας ε, ε, εκπροσωπεί πια τον ανάδοχο επιχειρηματία στην Κίνα. Έχουν δηλαδή συνεργασία στις διεθνείς αγορές. Η δεύτερη εμπειρία αφορά τον τουρισμό και έναν νέο επιχειρηματία, το Ιούκα Καταράκο που έκανε ανταλλαγή τετράμινη στην Ισπανία και έκτοτε επέκτηνε τις επαγγελματικέ του δραστηριότητες και στην Ισπανία. Τώρα δηλαδή έχει ε, ε, δραστηριότητες και στη Φιλανδία και στην Ισπανία σε στενή συνεργασία με τον ανάδοχο επιχειρηματία. Πριν τη δημόσια ακρόαση, πραγματοποιήσαμε μία έρευνα στους ενδιάμεσους, στις ενδιάμεσες οργανώσεις. Στείλαμε ερωτηματολόγιο σε όλους ε, όσοι έλαβα την πρόσκληση για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση του δικτύου το, το περασμένο Φεβρουαρίου και 42 μας απάντησαν. Είπαν ότι ε, αφιέρωνα μία με δύο ώρες τη μέρα στο πρόγραμμα αυτό οι ενδιάμεσες οργανώσεις για τις ανταλλαγές των επιχειρηματιών. Βέβαια το ποσοστό ποικίλει. Στην αρχή όταν κανείς πρωτομπαίνει στο πρόγραμμα αφιερώνει περισσότερες ώρες στην προώθηση του προγράμματος, στην ευαισθητοποίηση του κοινού, στο να γνωστοποιήσει το πρόγραμμα, αλλά από τη στιγμή που έχει μπει σε ρότα, βοηθούμε τους ε, επιχειρηματίες, αλλά η προώθηση του προγράμματος ε, στους ε, επόμενους κύκλους δεν είναι τόσο χρονοβόρα όσο στον αρχικό κύκλο. Εξαρτάται φυσικά και αυτό και από τους επιχειρηματίες. Θα ταξινομούσα τους νέους επιχειρηματίες, ε, τους, νέους επιχειρημα... τους νεαρούς επιχειρηματίες σε τρεις κατηγορίες. Έχουμε καταρχήν εκείνους που, είναι, που πραγματικά ανοίγουν θέλουν να ανοίξουν τη δική τους δουλειά, ξέρουν τι θέλουν, έχουν κατά νου συγκεκριμένους στόχους και αναζητούν τον τέλειο ανάδοχο για να, για να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους. Αυτοί δεν χρειάζονται και μεγάλη συνδρομή από τους ενδιάμεσους οργανισμούς. Η δεύτερη κατηγορία των νέων επιχειρηματιών είναι εκείνοι που έχουν ενθουσιασμό, αλλά θέλουν κάποια βοήθεια και στήριξη είτε στα προγράμματα δράσης, είτε στα επιχειρησιακά προγράμματα. Θέλουν βοήθεια λοιπόν και σε γλωσσικό επίπεδο όταν Υποβάλλω την αίτηση του προγράμματος για να έρθουν σε επαφή με τον ανάδοχο. Και έχουμε και την τρίτη κατηγορία, Του νέου επιχειρηματίε που περιμένουν ιδιαίτερη μεταχείριση. Εμείς επικεντρωνόμαστε κυρίω ε, στι δύο πρώτε κατηγορίες. Η τρίτη δεν είναι κατηγορία, δεν είναι γνήσιοι επιχειρηματίες, γιατί θα πρέπει από μόνοι τους να θέλουν να ξεκινήσουν ε, μια επιχείρηση. Η μεγαλύτερη πρόκληση του προγράμματος, όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα της έρευνας, είναι να προσελκύσουμε ανάδοχους επιχειρηματίες που εργάζονται αμυστή στο πρόγραμμα, εθελοντικά. Από τη στιγμή όμως που βρούμε τους αναδόχους, ε, αναλαμβάνουν στη συνέχεια περισσότερους νέους επιχειρηματίες. Δηλαδή, η αρχή είναι δύσκολη. Από τη στιγμή που κάποιος μπει στο πρόγραμμα ως ανάδοχος, μετά ευχαρίστως συνεχίζει τις ανταλλαγές. Επίσης δύσκολο θέμα ήταν και η αξιολόγηση των συνεπειών των ανταλλαγών ένα εξάμεινο μετά τις, αλλαγές, τις ανταλλαγές. Ο επιχειρηματίας ε, θα πρέπει να αποφασίσει πότε θα ξεκινήσει την επιχείρηση του αμέσως ή λίγο αργότερα μετά το πέρας της ανταλλαγής. Συνήθω 6, με 12 μήνες μετά την ανταλλαγή ο επιχειρηματίας ε, μπαίνει στα βαθιά και ξεκινάει τη δική του επιχείρηση. Ο προλαλή σα. αναφέρθηκε στην ανάγκη απλούστευση των διαδικασιών και αυτή είναι πρόκληση. Και έτοιμα και των ενδιαφερομένων. Και τα εργαλεία πληροφοριών και επικοινωνιών στον τομέα αυτό παρουσιάζουν κάποια τεχνικά προβλήματα που συνεχώς βελτιώνονται. Ήδη τον τελευταίο χρόνο είχαμε σημαντική πρόοδο. Παρ' όλα αυτά, μερικές επιχειρήσεις έχουν προβλήματα με τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών που χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν. Μερικοί μάλιστα εξαρτούνται πλήρως από, τους, από τις ενδιάμεσες οργανώσεις. Αυτές βοηθούν τους επιχειρηματίες να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση και να κάνουν και τις υπόλοιπες διατυπώσεις. Βέβαια, οι νέοι επιχειρηματίες που είναι και νεαροί είναι πολύ πιο εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και αντιμετωπίζουν πολύ πιο εύκολα τα τεχνικά προβλήματα. Τώρα, ποιες είναι οι υπόλοιπες προκλήσεις εκπρόσωποι των διάμεσων οργανώσεων αναφέρθηκαν στις, στους δημοσιονομικούς περιορισμούς και στις επιδοτήσεις για τους νέους επιχειρηματίες, γιατί δυστυχώς ε, δεν υπάρχουν πολλά κονδύλια, γι' αυτό και χρειάζεται να βάζουν ε, στο περίμενε τους νέους επιχειρηματίες ε, μέχρι ότου να εξασφαλίσουν τα κονδύλια. Επίσης πρέπει να εξηγήσουν στον ανάδοχο ότι δυστυχώς δεν μπορούν να δεν μπορούν να τους στείλουν αμέσως τον επιχειρηματή γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Επίσης έχουμε κάποιες ενδιάμεσες οργανώσεις που είναι κάπως παθητικές, δεν είναι και πολύ δραστήριες. Ή έχουμε τους νέους ερχόμενους, για τον πέμπτο κύκλο είχαμε νέες οργανώσεις ενδιάμεσες. Ξεκίνησαν από το Φεβρουάριο. Είναι η πρώτη σε επαφή με το πρόγραμμα, οπότε θα χρειαστούν λίγο χρόνο να εξοικειωθούν και με τις ε, διαδικασίες μέσω των υπολογιστών. Οπότε αυτοί που κάνουν τα ταιριάσματα αφιερώνουν κάποιο χρόνο στην κατάρτιση και των νέων ε, ενδιάμεσων οργανώσεων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο καθήκον τους και αυτές. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις ενδιάμεσες οργανώσεις να εφαρμόσουν το πρόγραμμα για τους νέους επιχειρηματίες πιο αποτελεσματικά. Καταρχήν με την απλούστευση της διαδικασίας ε, της ηλεκτρονικής υποβολής και καλύτερη συνεργασία των ενδιάμεσων οργανώσεων ε, και στο εσωτερικό μιας χώρας. Στη Φιλανδία έχουμε τρεις τέτοιες οργανώσεις με πολύ στενή δικτύωση και πολύ στενές επαφές. Οπότε έχουμε κοινά ανακοινωθέντα τύπου, κοινέ ε, εκστρατείε γνωστοποίηση ε, ενημερωτικέ, αλλά πάντα υπάρχει χώρο για βελτίωση τη συνεργασία. Επίση, η διαχείριση των κονδυλίων θα πρέπει να γίνει πιο αποκεντρωμένα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 10% το όριο και αυτό, αυτό εφαρμόζουμε. Εφόσον όμως έχουμε εταίρους που δεν έχουν αρκετές επιδόσεις, που δεν λαμβάνουν ε, αρκετές αιτήσει από νέου επιχειρηματίες, θα πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα μεταφοράς ε, των κονδυλίων προς εταίρους, ε, προς, προς διάμεσο που κατακλείζονται από αιτήσει νέων επιχειρηματιών και δεν έχουν αρκετό προϋπολογισμό. Θα πρέπει να υπάρχει μια ελαστικότητα για τη μεταφορά των επιδοτήσεων. Ποια είναι τα σημαντικότερα διδάγματα που αντλήσαμε από το πρόγραμμα. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ήθελα και εγώ να επισημάνω ότι μερικές φορές είναι παραπλανητικός ο τίτλος του προγράμματος, η ονομασία του προγράμματος. Για πολλούς το έρασμος ε, ε, προκαλεί τον άμεσο συνειρμό της ανταλλαγής των σπουδαστών. Και όταν μερικές φορές λέμε νέους επιχειρηματίες, πρόγραμμα για νέους επιχειρηματίες, μερικοί θεωρούν ότι το νέος αφορά την ηλικία, όχι στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Αλλά το νέος καλύπτει όχι μόνο την ηλικία, αλλά το, την επιχειρηματική δραστηριότητα. Νέο στη δουλειά, όχι νέο στα χρόνια κατά ανάγκη. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε τις ε, κοινέ προσπάθειες ε, των ε, διάμεσων οργανώσεων στις διάφορες αγορές. Θα πρέπει να γίνεται και τοπική πρόθεση του προγράμματος εθνικά με τη συνεργασία των τοπικών των, τοπικών ενδιάμεσων οργανώσεων. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε στενή συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων ενδιάμεσων οργανισμών. Εμείς είμαστε πανεπιστήμιο, αλλά μας βοήθησαν και ενώσεις ενδιάμεσων οργανισμών και ε, επιμελητήρια και μάλιστα μας βοήθησε και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων το παράρτημα του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιδιώκουμε σύσφυξη της συνεργασίας και με το δίκτυο αυτό. Όπως ακούσαμε, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ποιότητα, που είναι πολύ σημαντικό και αξιέπαινο στόχος του προγράμματος, όχι μόνο τώρα αλλά και για το μέλλον. Επίσης, έχουμε ειδικά προγράμματα τομεακά. Όταν κανείς υποβάλλει αίτηση για το πρόγραμμα Έρασμος για νέους επιχειρηματίες, η περιγραφή ε, το, της επαγγελματικής δραστηριότητας, στην περίπτωσή μας αφορά τον τουρισμό, αλλά δεχόμαστε αιτήσεις και από άλλους επιχειρηματικούς κλάδους. Για εύλογους λόγους όμως, εμείς διαλέξαμε τον τουρισμό και επικεντρωνόμαστε στον τουρισμό. Οπότε ανακύπτει το ερώτημα. Έχουμε δικαίωμα να περιοριζόμαστε σε ένα και μόνο κλάδο. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στους νέους κύκλους ε, λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη επίδοση των διάμεσων οργανώσεων. Γιατί, όπως σας είπα, υπάρχουν και παθητικές και πιο δραστήριες οργανώσεις οι επιδόσεις τους διαφέρουν στην επαφή τους με το πρόγραμμα και το, τους επιχειρηματίες. Η πείρα λοιπόν της διάμεσης οργάνωσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και οι επιδόσεις της όταν υποβάλλονται αιτήσει για τους νέους κύκλους. Επίσης προτάθηκαν πιο μεγάλες περίοδοι εφαρμογής. Για τον έκτο κύκλο είναι 24 μήνες. Στο παρελθόν ήταν 21 μήνες η διάρκεια τιμών ε, ακόμη μεγαλύτερες περίοδους, 3 με 5 χρόνια, ώστε να εξασφαλιστεί μια συνέχεια με τους επιχειρηματίες και τους στόχους. Τώρα, γεωγραφική διεύρυνση. Παρόμοιες πρωτοβουλίες είχαμε και στο παρελθόν, όπως ανταλλαγές Ευρωπαϊκής Ένωσης Βραζιλίας. Μάλιστα σκεφτήκαμε να υποβάλουμε αίτηση και για το πρόγραμμα αυτό, αλλά θεωρήσαμε ότι οι επιχορηγής αυτού του προγράμματος περιοριζόταν σε 250 ευρώ το μήνα. Αυτό θα μας σκότωνε πραγματικά γιατί με τόσο μικρή επιδότηση δεν είναι πολύ δελεαστική πρόταση για τους νέους επιχειρηματίες. Πάντως ε, υπάρχει μια, ένας πολλαπλασιασμός των πρωτοβουλειών αυτών. Εγώ ασχολήθηκα με την προώθηση του προγράμματος στην Νοτιοανατολική Ασία και το Βιετνάμ. Και εκεί υπάρχει ενδιαφέρον για τέτοιες πρωτοβουλίες. Και μάλιστα ήρθαν κάποιοι εκπρόσωποι των χωρών αυτών που είπαν ότι θα εξετάσουν και θα διερευνήσουν τη δυνατότητα εφαρμογής ε, τέτοιων προγραμμάτων και στο δικό τους έδαφος. Αυτά λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Τέτοιου είδους προγράμματα είναι πολύ χρήσιμα γιατί πραγματικά έχουν απτά αποτελέσματα και τα χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ. Very much. Uh, I'm happy that you Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιβεβαιώνετε ότι πραγματικά η Ευρώπη είναι στην ηγεσία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματικά δημιουργήσε ένα πρόγραμμα το οποίο συμβάλλει στην ε, μείωση της αναργίας. Νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τη συζήτηση. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσεις, ε, παρατηρήσεις από τους βουλευτές. Έχετε το λόγο. Η κυρία Χέρτσοκ, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Ρούμπεχ. Φαντάζεται κανείς ότι ε, όταν κάποιος κάθεται εδώ για δύο ώρες και ακούει τις παρουσιάσεις, κάτι θέλει να πει. Χαίρομαι που για πρώτη φορά προσθέσαμε μία παράγραφο για το Erasmus για τους νέους επιχειρηματίες στο Small Business Act και στη σχετική έκθεση για την οποία ήμουν εισηγήτρια. Και μετά ακολούθησε η πρωτοβουλία του κύριου Ρίμπιχ, την οποία προσυπέγραψα και οδήγησε στο επιτυχές πληθυκό πρόγραμμα. Είναι σημαντικό να το ξέρουν οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Προπολογισμών ότι πρόκειται για ένα από τα πιο επιτυχή προγράμματα με απτά, απτά αποτελέσματα και μεγάλη επιτυχία. Και εγώ μαζί με εσά ε, παρευρέθησα σε μία εκδήλωση όπου γνωρίσαμε τους επιχειρηματίες αυτές. Ένας Ιταλός ε, παραγωγός ε, παγωτού από τη Λούκα ήρθε σε επαφή με Ισπανό επιχειρηματία από τη Βαρκελόνη και τελικά μαζί συνεργάστηκαν και δημιούργησαν πραγματικά εκπληκτικά αποτελέσματα για τα εστιατόρια. Είναι πραγματικά ενδεικτικό της επιτυχίας του προγράμματος. Να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του κ. Βάινμπεργκερ, πώς μπορούμε να προωθήσουμε καλύτερα το πρόγραμμα αυτό από κοινού με την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Είναι εμβληματικό πρόγραμμα αυτό το ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου. Και γι' αυτό λοιπόν ε, πιστεύω ότι είναι το καταξοχήν πρόγραμμα το Εράσμου για τους νέους επιχειρηματίες. Όπως είπε και ο κύριος Σαμπροτζίνη. πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποδοτικοί. Καταρχάς να συνεχίσουμε να προωθούμε το πρόγραμμα, αλλά και κατά δεύτερον ένας νέος επιχειρηματός, ε, επιχειρηματίας να μεταδίδει, αν θέλετε, τα φώτα τους άλλων νέων επιχειρηματιών Κάτι άλλο το υπογραμμίσω, το οποίο δεν ακούσουμε επαρκώς. Ότι πρόκειται για μια οργάνωση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, των νέων επιχειρηματιών ανεξάρτητος ηλικία. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους πρόθεση λοιπόν του προγράμματος αυτού από το πλευρά του Κοινοβουλίου. Να μην μείνει απ' έξω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθότι στο Κοινοβούλιο ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό. Παρά το γεγονός ότι μας συμβούλευσαν και μας βοήθησαν πολύ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα ο κ. Βάινμπεργκερ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω πρέπει να προβληθεί στο πλαίσιο αυτό. και να κοιτάξουμε και τις άλλες επιτροπές, γιατί προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα το πολιτισμικό, στον τομέα το ψηφιακό. Και ίσως οι συνάδελφοι στις άλλες επιτροπές να μην γνωρίζουν το πρόγραμμα αυτό τόσο σε βάθος όσο στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Άρα, συνοψίσοντας, πολύ καλή δουλειά, πολύ σημαντική επιτυχία βρείτε νέους επιχειρηματίε από τις χώρες σας για να μοιραστούν και αυτή την επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρία Έρτσοκ, λέει ο κύριος Ρούμπιχ. Αυτό καταδεικνύει ότι τα πρωτικά μας προγράμματα στέφονται πραγματικά με επιτυχία. Ευχαριστώ και τους συντονιστές που μας υποστήριξαν σε κάθε περίπτωση. Η κυρία Βέρτμαν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μα για τα προγράμματα αυτά, για το πρόγραμμα αυτό. Δύο ερωτήσει να κάνω προ τον κύριο Βάινμπεργκ, αν μου επιτρέπετε, ποσοστιαία αναχώρα ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας. Ωραία, διεξάγεται το πρόγραμμα. Αλλά ποιοι επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται ως επιχειρηματίες και μετά από πέντε χρόνια. Για να δούμε πώς μπορούμε να επεκτείνουμε ενδεχομένω το πρόγραμμα και να δούμε και ποιες είναι οι διαφορές αναχώρα. Δεύτερη ερώτηση τώρα. Υπάρχουν πρωτοβουλίες, υπάρχουν σκέψεις για το κατά πόσον αυτό το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί στις ε, χώρες που αντιμετωπίζουν την κρίση, την Ελλάδα, την Πορτογαλία. Έχουμε μεγάλο, τεράστιο ποσοστό ανεργίας στους νέους και έτσι θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση, να δώσουμε, αν θέλετε, ε, ένα λόγο και ένα κίνητρο να ενθουσιαστούν οι νέοι και σε αυτές τις χώρες και να δραστηριοποιηθούν. Ευχαριστώ, κυρία Τρίπελ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα σας προκαλέσει έκπληξη το γεγονό ότι λίγο πολύ οι ερωτήσει μου θα κινηθούν προ την ίδια κατεύθυνση όπω και οι δύο προλαλήσασε. Είναι πάρα πολύ καλό το ότι βλέπουμε σε κάποιο βαθμό την επιτυχία του προγράμματος, όπως και το πρόγραμμα Εράσμου για τους φοιτητέ. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η αρχή ανταλλαγής ε, φοιτητών, επιχειρηματιών, νέων ανθρώπων, προκειμένου να έρθουν σε επαφή από τον κόσμο, αν θέλετε, της εκπαίδευσης με τον κόσμο των επιχειρήσεων. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της ενεργείας των νέων. Να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο όλο front-loading θα προσπαθήσετε να κάνετε πιο πολλά σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα αυτό. Γιατί έχει αποδεχτεί επιτυχές και σε ό,τι αφορά λοιπόν τη χρηματοδότηση και σε ό,τι αφορά την προετοιμασία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι ακριβώς λοιπόν θα εφαρμόσετε και θα χρησιμοποιήσετε. Μιλήσατε και για την καλύτερη διαφήμιση και προώθηση του προγράμματος. Τι προτείνετε. Τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε και μπορούμε να κάνουμε παραπάνω στην παρούσα χρονική συγκυρία. Προφανώς υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη επιτυχία και άλλες που δεν υποστηρίζουν το πρόγραμμα αυτό στο ίδιο βαθμό. Και τι μπορούμε να κάνουμε, όπως είπε και η κυρία Βέρτημα, στις χώρες που αντιμετωπίζουν πιο έντονα την κρίση. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανείς άλλος να ζητάει τη λόγο. Εγώ ως εισηγητής θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι ποσό χρειάζεται προκειμένου στο 2014 να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με επιτυχία το πρόγραμμα. Κύριε Βάινμπεργκερ, αν θέλετε να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολλές και ενδιαφέρουσες οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις. Όπως σας είπα, προετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή την ανασκόπηση των τελευταίων πέντε ετών, προσπαθώντας να δούμε ποιοι παράγοντες βοηθάν και ποιοι περιορίζουν. Οι περισσότερες λοιπόν ερωτήσεις θα απαντηθούν μόνο εκ των υστέρων, ιδιαίτερα γιατί πέντε χρόνια μετά που είναι η μακροχρόνια προσέγγιση δεν έχουμε ακόμα κανέναν. Κάποιοι έχουν μια τριετία και σε αυτούς απευθυνθούμε στην αξιολόγηση για να τους ρωτήσουμε ποιος ήταν ο αντίκτυπος για αυτούς. κάναμε μια ανάλυση αντικτύπου όταν ετοιμάζαμε την νομική βάση του προγράμματος και ήταν σαφές ότι ο οικονομικός αντίκτυπος μπορεί να είναι τεράστιος η ανάλυση, ήταν σαφής, έλεγε. Αν δημιουργούνται δύο θέσεις εργασίας με κάθε startup και μέσω διεθνών συνεργασιών ή καινοτόμων ε, δραστηριοτήτων θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Η απόδειξη, ήταν... η απόδειξη είναι το δύσκολο, αλλά ο αντίκτυπο εν δυνάμει είναι τεράστιο. Για τις χώρες να απαντήσω τώρα. Υπάρχει μία στρέβλωση. Οι 40% των σχέσεων είναι σε δύο χώρες, που είναι και οι δύο χώρες κρίσης, τα Ισπανία και η Ιταλία. Αλλά και εκεί υπάρχει επιτυχία. Οι ανταλλαγέ λοιπόν είναι πολύ επιτυχείς. Η κύρια παρατήρηση είναι εξαρτάται πολύ από το αν έχουμε ενδιάμεσους οργανισμούς. και ο κίνδυνος είναι να μην υπάρξει η εικόνα της επιτυχίας. Τώρα, καλη Σημαντική πρόοφηση, Αλλά είναι πρόοφηση όταν έχουμε πολλές αιτήσει και καμία ε, ε, και καμία συνέχεια γιατί δεν έχουμε επαρκή, κονδύλια στον προπολογισμό. Από 700 πήγαμε σε 2.000 αιτήσει που, είχαν, που είχαν γίνει δεκτές. Για τα επόμενα τρία χρόνια δηλαδή, αν θέλετε, έχουμε κλείσει. Χωρίς περισσότερα κονδύλια δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και η προώθηση είναι, θα ήταν λάθος. Η προώθηση για να αποκτήσεις νέους επιχειρηματίες που μετά δεν μπορείς να ικανοποιήσεις δεν είναι παραγωγικό. Τώρα, επέκταση σε άλλες χώρες. Μα περάσαμε ήδη σε 37 χώρες, όλες τις χώρες με τις οποίες έχουμε συνεργασία. Ευχαριστώ και την ερώτηση παρεμπιπτόντος από τη Φινανδία. Μία με δύο ώρες δεν είναι αρκετή. Δεν καλύπτει την κρίσιμη μάζα. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε αρκετούς φορείς, ενδιάμεσους φορείς που τρώνε, που δαπανούν 5-6 ώρες την ημέρα για να δουλε, δουλεύονται στο πρόγραμμα, γιατί έτσι γίνεσαι παραγωγικός αν θέλουμε να έχουμε κέρδη παραγωγικότητας. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να κάνουμε περαιτέρω προβολή και πρόθεση, αλλά να μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Ε, προφανώς η ενεργεία των νέων πρέπει να είναι βασικός στόχος στο πλαίσιο αυτό και αυτό που είδαμε είναι η δράση ανεργίας, η δράση για την ανεργία ούτως ώστε ο κόσμος να αποκτήσει τη δυνατότητα να ξεκινήσει μόνος του μια επιχείρηση ήδη έχουν γίνει την τελευταία οκταετία, δεκαετία. Σε πολλές περιπτώσεις ήταν επιτυχής. Διαπιστώνουμε ωστόσο ότι για να επιβιώσουν τα πρώτα δύο χρόνια είναι κρίσιμη η καλή προετοιμασία. Και εδώ βοηθά το πρόγραμμα, γιατί μειώνει με καλή προετοιμασία το την πιθανότητα αποτυχίας. Πρέπει απλά με τη σωστή συμπεριφορά να ξεπεράσουμε τα προβλήματα κλίμακας. Αλλά από την άλλη, μην ξεχνάτε ότι και εμείς έχουμε ε, ε, περιορισμούς στο ανθρώπινο δυναμικό μας. Λίγους ανθρώπους έχουμε. Έχουμε υποχρεώσεις βάσει του χρηματοοικονομικού κανονισμού που απαιτεί μεγάλη γραφειοκρατική επιβάρυνση και στην Επιτροπή, για να σας πω την αλήθεια, δεν έχουμε ανθρώπινους πόρους αρκετούς για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν ή να αντιμετωπιστούν όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα. Έχουμε προβλήματα ε, κίνηση ε, κλιμάκας, όχι πια προβλήματα αύξησης. Τέθηκε το ερώτημα της εξειδίκευσης. Καλή είναι η εξειδίκευση, αλλά όταν έχεις μικρό προπολογισμό, θέλουμε κάθε ενδιάμεσο οργανισμό να δραστηριοποιείται 5 με 6 μήνες, ε, ώρες την ημέρα, άρα να πληρώνεται. Δεν μπορούμε να διευρύνουμε λοιπόν το στόχο μας, το στόχο μας ούτε να μπούμε σε όλους τους τομείς. Μπαίνουμε λοιπόν σε γενικευμένη προσέγγιση προς το παρόν. Τώρα για την κρίσιμη ερώτηση. Ποιο είναι ο σωστό προπολογισμό. Αφενό, όπως είπα, έχουμε αιτήσει για 20, για 35.000 ενώ μπορούμε να καλύψουμε 5.000 θέσεις. Συνολικά μπορεί να έχουμε προγράμματα 17-18.000 ευρώ. Για το 13 μας λείπουν άλλα τόσα για να χρηματοδοτήσουμε το ενδιαφέρον που, αυξάθηκε, που αυξήθηκε. Έχουν περισσότερες προτάσεις σε σχέση με το παρελθόν. Όταν μιλάμε όμως για 10.000 επιχειρηματίες κάθε χρόνο που είναι ο στόχος για το, 20, για το 2020, Είπε ο κύριο Αμπρουτσίνη ότι μπορούμε να μειώσουμε το κόστο κόστος επιχειρηματία. Σωστό. Αλλά υπάρχουν όρια. Αν το κόστο που δίνεται στου επιχειρηματιε είναι 4 με 5.000 ευρώ και θέλει να προσλάβει προσωπικό και του πληρώσει για να δουλεύουν σχεδόν full time για το project, ε, πόση μείωση μπορεί να έχει, και να πούμε λοιπόν ότι το 7.000 είναι καλό νούμερο, το θέμα είναι θέμα αριθμητική. 7.000 επί 10.000 επιχειρηματίες είναι 70 εκατομμύρια. Ενώ εμείς έχουμε 50 για 7 χρόνια. Δεν μιλάμε για 10-20% λοιπόν διαφορά. Θα πρέπει να αυξήσουμε και τους ανθρώπινους πόρους που διατίθενται στην Επιτροπή. Πολλά γίνονται μέσω της εξωτερικής ανάθεσης. Αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ. Δεν μπορεί να γίνει αυτή Άλλοι ζητούν μείωση, τα, τα κράτη μέσα ζητούν μείωση 50% του ε, προσωπικού της Επιτροπής. Το κρίσιμο στοιχείο είναι να κρατήσουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Κυρία Μπρίνκεβιτσούτη, κυρία Γκλέσλερ και μετά θα απαντήσετε. Well, uh, just, Ευχαριστώ. Λίγα σχόλια για τα νέα στοιχεία από τη συμπερίληψη πρόσφατα το Φεβρουάριο του έρασμος για τους νέους ε, επιχειρηματίες ε, στο κόσμο. Ε, υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες στο, στο κρατικό επιμελητήριο που είναι το σημείο επαφής για να βοηθήσουν τους νέους επιχειρηματίες να αντιληφθούν πώς λειτουργεί η αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουν να αντισταθούν στις πιέσεις αγοράς και να βρουν καλές καλές λύσεις. Είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα αυτό και πιστεύω ότι θα προσελκύσει ζωηρό ενδιαφέρον. Βρισκόμαστε σε φάση τώρα της ε, ενημέρωσης ε, και της εκπαίδευσης. Και εγώ ως Ευρωβουλευτής θα προσπαθήσω να βοηθήσω τις αρμόδιες υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ε, συνδράμουν το σημείο επαφή στην Κροατία που είναι το κρατικό εμπορικό επιμελητήριο για να βελτιωθεί η εφαρμογή του προγράμματος και εκεί. Κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την ελαστικότητα για τη μεταφορά των κονδυλίων, θα ήθελα να ρωτήσω ε, ποια άρθρα του προϋπολογισμού του, για το δημοσιονομικό θέμα εμποδίζουν τη μεταφορά των κονδυλίων. Κύριε Γκαρίγα, και εγώ έχω μία πολύ απλή ερώτηση προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποιο είναι το ποσοστό εκτέλεσης του προγράμματος Έρασμος ε, για τους νέους επιχειρηματίες από την έναρξη του προγράμματος μέχρι τώρα Η ερώτηση είναι το ότι ποιε είναι οι δυνατότητε στα πλαίσια του προπολογισμού του 2014. Τι κονδύλια χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση του 2014. Ο συνάδελφο Ευχαριστώ για τα σχόλια από την Κροατία. Σίγουρα οι διάμεσε οργανώσει ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ και ελπίζω να αρχίσουν να λειτουργούν το συντομότερο δυνατό και στην Κροατία. Σε ό,τι αφορά το άρθρο του δημοσιονομικού κανονισμού, ευχαριστώ για την ερώτηση, πολύ συγκεκριμένη κυρία Γκρέσλε, αλλά δεν θυμάμαι απ' έξω. Θα το κοιτάξω και θα σας ε, στείλω γραπτό στην απάντηση. Ναι, αλλά θα με ενδιαφέρε να μου απαντήσετε. σα παρακαλώ, μην ε, μου βλέπετε ότι θα στείλετε μόνο ένα... Μην καθυστερήσετε να μου στείλετε το email. Ναι, ναι, ναι, θέλετε άμεσα τι πληροφορίε αυτά με email. Δεν σα υπόσχομαι τίποτα, κυρία Γκρέσλε. Σε ό,τι αφορά το ποστό εκτέλεση. Τα πρώτα χρόνια εφαρμογή ήταν χαμηλό το ποσοστό εκτέλεση του Εράσμου δεν ήταν και πολύ πεπειραμένε οι διάμεσες οργανώσεις, ε, δεν ήταν πολύ γνωστό το πρόγραμμα. Πάντω μα ενδιαφέρουν κυρίω τα αποτελέσματα. Αν μια διάμεση οργάνωση δεν είχε καλέ επιδόσεις, δεν ανταπεξήλθε στο έργο τη. και μόνο το 10% των σχέσεων προώθησε, σίγουρα θα λάβει πλήρη χρηματοδότηση. Δεν θα λάβει το 100% της χρηματοδότησης. Τα πρώτα δύο χρόνια το ποσοστό εκτέλεση ήταν πολύ χαμηλό γύρω στο 25 με 30% σε ό,τι αφορά τις πληρώσεις, τις πιστώσεις πληρωμών. Σε ό,τι αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων, υπήρξε αύξηση. Ήταν σημαντικό το ποσοστό, αλλά σε ό,τι αφορά τις πληρωμές ήταν χαμηλό το ποσοστό εκτέλεσης. Αλλά για τις πιστώσεις ανάλυσης υποχρεώσεων δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, ξεπερνούσαμε και το πρόγραμμα 120%. Τώρα για το 2014 οι προβλέψεις είναι, είναι 17 εκατομμύρια. Ε, τα τελευταία χρόνια είχαμε συνεχίσει μειώσει. θα έλεγα 20 εκατομμύρια αισιόδοξη πρόβλεψη για να διευρυθεί το πρόγραμμα όσο γίνεται περισσότερο, να περάσουμε από τα 17 στα 20. Σας ευχαριστώ ο εισηγητής για το θέμα αυτό. Θα ήθελα κυρίως να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες στις σημερινές ακροάσεις που μας βοήθησαν στην εφαρμογή του προγράμματος το οποίο ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να καταστεί ένα πρόγραμμα με ιδιαίτερη επιτυχία και πραγματικά η Ευρώπη να βρίσκεται στην κορυφή αν θέλετε της ε, καινοτομία σε ό,τι αφορά αυτό το πρόγραμμα, το οποίο καταπολεμά και την ανεργία, δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους σας ε, όσοι συμμετείχατε σε αυτή τη διαδικασία και σας ε, παρακαλώ να συνεχίσετε να υποστηρίζετε το πρόγραμμα αυτό. Και δίνω την Προεδρία τώρα στη συνάδελφο Γιούτα Χάουκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα περνάμε πάρα αυτά ένα άλλο θέμα το οποίο είναι ασφαλώς εξίσου σημαντικό και χρήσιμο. Οι νέοι επιχειρηματίες έχουν αποδείξει ότι σίγουρα μπορούν να τηρούν το χρονοδιάγραμμα. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερως για αυτό. Και τώρα περνάμε στην ετήσια συνεδρίαση Μιλάμε πάντα για τους οργανισμούς παρά το γεγονός ότι και εκεί έχει καθιερωθεί το μέσο της Τρόικας, το εργαλείο της Τρόικας. Έχουμε όλο και πιο, πολύ, πιο πολλούς ε, αποκεντρωμένους οργανισμούς. Προκειμένου λοιπόν να μην ε, χρειαζόμαστε κάθε φορά δύο-τρεις μέρες για να τους ακούμε όλους εδώ. Εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα υπάρχει μια τρόικα και σε αυτό το πλαίσιο. Και αυτή η τρόικα λοιπόν εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει αυτούς τους οργανισμούς και συζητά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτά που απασχολούν όλους τους οργανισμούς. Φύγει και τα προβληματικά σημεία. Ασφαλώς είναι πάντα καλό να μαθαίνουμε το τι πηγαίνει καλά και τι είναι ιδιαιτερός θετικό, αλλά μιας και έχουμε περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μας, θα σας δώσουμε το λόγο, θα συζητήσουμε τον προπολογισμό, το σχέδιο προπολογισμού που μας ε, διαβίβασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορά ασφαλώς και τον προϋπολογισμό για τους οργανισμούς και παράλληλα θέλουμε να συζητήσουμε και αυτά τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά το προσωπικό των οργανισμών. Προτείνει τα προβλήματα που μας προκαλεί, πώς να το πω. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε ενδεχομένω και να μην το προεξοφλήσω. Να δούμε ποια είναι η αντίδραση των ε, οργανισμών. Ποιοι θα μιλήσουν, ο διευθυντής ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνδρομικών Οργανώσεων, κύριε Μασλίκ, ελπίζω σωστά να πρόφερα το όνομά σας. Μόρταν Κέρουμ, Διευθυντή. του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από τη Βιέννη. Ελπίζω να μην είναι εδώ μαζί μας σήμερα επειδή θεωρεί ότι πλήττονται τα δικαιώματα των ίδιων των οργανισμών. Ανδρέα Αμών, αναπληρωτής ε, διευθυντής του ECDC του Ευρωπαϊκού Κέντρου. Καλώς ορίσατε. Δίνω το λόγο στον κύριο Φρενσίκ για να μας κάνει την εισήγηση του. Σας ευχαριστώ. Ως Βέλγος προφέρεται διαφορετικά το όνομά μου. Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να κάνουμε συζητήσεις για τον υπολογισμό του 14 και την παρουσίαση της κοινής προσέγγισης. Σας δοκιμάσαμε ένα κείμενο, όπως συνήθως έχουμε μια πλήρη εικόνα, παρουσιάζει μια πλήρη εικόνα της κατάστασης και τις επιπτώσεις της, των αρνητικών επιπτώσεων του προπολογισμού στις διάφορες υπηρεσίε. Πριν δύο εβδομάδες είδαμε την πρόταση της Επιτροπής για τον προπολογισμό του 2014 και τώρα προσπαθούν οι υπηρεσίε μας να βρουν καλύτερες πληροφορίες, περισσότερες πληροφορίες για το τι κρύβεται πίσω από αυτό. Ωστόσο πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σήμερα στο συμπέρασμα ότι για το 14 και μετά η εικόνα είναι σκοτεινή. Η μείωση σε προσωπικό και κονδύλια πάει παραπέρα από αυτό που αναμενόταν. Μερικές υπηρεσίες για παράδειγμα που τον περασμένο Δεκέμβριο είχαν θεωρηθεί ως νέες κατηγορίες υπηρεσιών για το 2014 και έπρεπε να προχωρήσουμε με ταχύτερους ρυθμούς, βλέπουν περικοπές. Εμείς προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την Επιτροπή για να αντιμετωπίσουμε ενιαίο πακέτο ως ενιαίο πακέτο της υπηρεσίας, αλλά αυτό σημαίνει ότι όταν ένας οργανισμός παίρνει επιπρόσθετους πόρους για να καλύψει τις υποχρεώσεις του, τότε αυτόματα οι πόροι των άλλων περικόπτονται. Από την άλλη πλευρά ωστόσο, ε, δεν αλλάζουν τα καθήκοντά του. Ο διαλόγος είναι ότι οι περισσότερε υπηρεσίε έχουν περικοπεί 2 ή και περισσότερο τη 100 του 14. Μέσα στα θεσμικά όργανα, στην κατηγορία 5, δεν υπάρχει μηχανισμό αντισταθμίσης και αν ένα όργανο υποστεί μείωση κατά λιγότερο από 1% η αύξηση των δαπανών του, δεν σημαίνει ότι τα άλλα όργανα πρέπει να μειώσουν τις ε, δαπάνες τους. Ξέρετε ότι μικρές δομές όπως ο διαμεσολαβητής, ο EDPS ε, δεν είχαν περικοπές, ενώ άλλες μικρές υπηρεσίες όπως όσας κλπ. είχαν περικοπή μεγαλύτερη του 2%. Αυτό σημαίνει ότι οι προτάσεις της Επιτροπής οδηγούν σε διαφοροποιημένη αντιμετώπιση των υπηρεσιών σε σχέση με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Θα, θα θέλαμε μια πιο συνεκτική προσέγγιση των υπηρεσιών. Ε, αφετηρία θα πρέπει να είναι τι περιμένουν από τις υπηρεσίες αυτές τα όργανα της Ένωσης. Ξέρουμε σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχει εξοικονόμηση λόγω του ότι η δουλειά γίνεται μία και όχι 28 φορές. Να τονίσω δύο παραδείγματα που βλέπετε στη θέση μας. Πρώτον, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης. Οι υπολογισμοί εκεί είναι ότι πέραν του 2% περικοπές η, η μείωση θα οδηγήσει σε περαιτέρω 7% μείωση του προσωπικού. Στο κέντρο μετάφρασης η περικοπή έγινε, είναι 4% φέτο και αυτό είναι ο λόγο τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπηρεσία αποφάσισε να μην γίνουν περαιτέρω περικοπές το 2014. Ωστόσο η Επίτροπη πρότεινε περαιτέρω περικοπή 1,5% παρότι το κέντρο αυτό χρηματοδοτείται απόλυτα. Ένα σημαντικό σημείο λαμβάνοντας υπόψη και την άφηξη της κρατικής γλώσσας. Όταν γράψαμε στο Κοινοβούλιο στην επιστολή της 29ης Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος Σούλτς τόνισε ότι το Κοινοβούλιο είχε πάντα την άποψη ότι τα καθήκοντα των υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από πόρους ό,τι αφορά το προσωπικό και τη χρηματοδότηση. Συμφωνούμε με την δήλωση του κ. Σούλτς τα παραδείγματα ωστόσο που σας δίνουμε δείχνουμε ότι το σχέδιο υπολογισμού έχει άλλη γλώσσα. Ξέρετε ότι οι υπηρεσίες έχουν στόχο να παράσχουν τα μέτρα, τις αρμοδιότητες που τους ζητείτε να γίνουν σε, κατα, σε περίοδους κακής οικονομικής συγκυρίας. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να υπάρχουν σαφείς και με διαφάνεια δραστηριότητες. η επίδοση των υπηρεσιών στο πλαίσιο αυτό είναι θετική. Πέραν αυτών αυξήθηκε και η συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών για να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της δουλειά μας. Πολλά παραδείγματα μπορούμε να σας δώσουμε. Δείχνουμε με τον τρόπο αυτό ότι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το καλύτερο δυνατό τρόπο την λειτουργία των υπηρεσιών και τα αποτελέσματα που έχουμε, αλλά βεβαίως υπάρχουν κάποια όρια διότι αυτό που μπορεί να πετύχουμε για τη μείωση του κόστους και των overhead είναι περιορισμένη. Είναι απογοητευτικό να βλέπεις ότι παρά τις, ε, τα καλά λόγια για την ανάγκη απλοποίησης κλπ. και λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, παρά τα αυτά έλεγα, ο νέος κανονισμός προσωπικού πηγαίνει στην ανάποδη κατάσταση. Δηλαδή αυξάνει το δημοσιονομικό βάρος των επιχειρήσεων και το συνολικό κόστος τους. Κάτι που έχει σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Στην τελευταία συνάντηση πέρσι, ο συνάδελφος που ήταν τότε πρόεδρος του δικτύου σας είχε ενημερώσει ότι ο μόνος ότι μία υπηρεσία από όλες δεν θα μπορούσαν με βάση τον υπολογισμό να τηρήσουν τις ε, υποχρεώσεις τους, αλλά μπορώ να σας πω φέτος ότι οι περισσότεροι, όλοι οι οργανισμοί στην ίδια κατάσταση βρίσκονται και θα πρέπει η Επιτροπή να επανεξετάσει τις αλλαγές στην ε, κατάσταση. Εφόσον η Δημοσιονομική Υπηρεχή πιστεύει ότι ο ρυθμός του προσωπικού και του προϋπολογισμού των υπηρεσιών πρέπει να μειωθεί, θα πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα στα διοικητικά συμβούλια για τα προγράμματα εργασία του 2014. Γιατί μία από τι δυσκολίε είναι ότι ενώ περικόπτονται οι προπολογισμοί, ξεκινά, αυξάνονται μάλλον τα καθήκοντα και κάθε φορά που η υπηρεσία κάνει μία πρόταση αναβολή, μείωση ή καθυστέρηση δραστηριοτήτων, αυτόματα η απάντηση είναι όχι, αυτό είναι προτεραιότητα. Αν όλες οι δραστηριότητες είναι προτεραιότητα, πώς μπορείς να προτεραιοποιήσεις τις προτεραιότητες. Ξέρουμε τι μας ζητείτε, αλλά πραγματικά είναι δύσκολο. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι ανησυχίες για τον προπολογισμό του επόμενου έτου. Οι αναπροσαρμογέ των μισθών, η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών σχολείων, που για κάποιε υπηρεσίε είναι σημαντικό, που περιγράφονται στην θέση που σα έχουμε παρουσιάσει. Δεν θα μπω περαιτέρω σε λεπτομέρειε. Είχα Συναντήσεις στην ε, συνάντηση της διαχείρισης για την ε, σύγκρουση συμφερόντων όπου η κυρία Γιάλα Σέντερ, εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου, είχε συστήσει στο Κοινοβούλιο υπήρχε μάλλον μια τάση αύξησης τη εξωτερική ανάθεσης δημιουργώντα μεγαλύτερα προβλήματα σύγκρουση συμφερόντων. Εμεί συμφωνούμε με την άποψη αυτή, ξέρουμε πολύ καλά Ξέρετε πολύ καλά έχουμε αυτό το θέμα της διαχείρισης των, ε, της σύγκρουσης συμφερόντων και, των και της ανεξαρτησίας της δομής. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι το προσωπικό του 2014 δεν θα πρέπει να ξεπεράσει το όριο αυτό. Η μεγαλύτερη ανησυχία μας είναι το πολιετές δημοσιονομικό πρέσιο. αντί να είναι χρήσιμο εργαλείο προγραμματισμού γίνεται ένα είδος Ζουλομάνδια Η απόκληση μεταξύ των αναγκών των υπηρεσιών και των πόρων τους αυξάνεται κάθε χρόνο, οδηγώντας σε αποδιοργάνωση των υπηρεσιών. Να πω και δύο λόγια ακόμα για την κοινή προσέγγιση και το roadmap της Επιτροπής. Όπως ξέρετε, το roadmap περιλαμβάνει 90 δράσεις που εμπλέκονται στην υλοποίηση όλων των περισσότερων από αυτές, έμεσα ή άμεσα. Αυτό το κάνουμε διότι πιστεύουμε ότι πολλά χρήσιμα πράγματα μπορεί να, προσέ... να προκύψουν από αυτή τη μακρά διαδικασία, αλλά απαιτεί και μέτρα και προσοχή. Η δουλειά του roadmap γίνεται σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και θέλω να τονίσω την στενή συνεργασία που έχουμε μεταξύ ε, υπηρεσιών και γενικής γραμματείας της ε, Επιτροπής. Ωστόσο υπάρχουν ανησυχίες για τη χρήση των μοντέλων που, παρουσιάζει, που παρουσιάζουν οι δομές αυτές. Δεν υπάρχει επαρκής δρόμος για να ληφθεί υπόψη ο ειδικός χαρακτήρας των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Σήμερα έχουν, υπάρχουν τέσσερις προτάσεις που έχουν γίνει και περιλαμβάνουν σημαντικά θέματα για την κοινή προσέγγιση. Οι υπηρεσίες θα ήθελαν να ξεκινήσουν ένα διάλογο με το Κοινοβούλιο για θέματα διακυβέρνησης και δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι αυτό δεν είναι εφικτό πάντα. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου τονίζει ότι αναγνωρίζει το Κοινοβούλιο τη σημασία των ε, υπηρεσιών και αυτό έχει αναπτυχθεί σαφώς. Νομίζω ότι Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει και καλύτερη συνοχή με τις υπηρεσίες. Έχω δίπλα μου τον κύριο Μόρτον Κέρμα από, την ΕΦΑΡ, από τη ΦΡΑ που είναι και πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Υπηρεσιών του χρόνου. Θα το κάνει παρότι θα χρειαστεί να μειώσει κατά 4% το προσωπικό του του χρόνου. Να σας πω ότι με χαρά Είμαστε σε διάλογο μαζί σας και με το Κοινοβούλιο και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε σε μόνιμη βάση την ποιότητα της διαχείρισης και τα παραδοτέα των υπηρεσιών μας. Τώρα όμως πραγματικά βρισκόμαστε σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Οι προοπτικές για το μέλλον δεν βοηθούν να έχουμε μια, μια αισιόδοξη προσέγγιση ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στο, στους συναδέλφους αν έχουν κάτι ακόμα να προσθέσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω και εγώ ότι καλύτερα θα ήταν να ακούσουμε πρώτα και τους τρεις ομιλητές. Και μετά να ξεκινήσουμε τον διάλογο με τους συνάδελφους. Ο κύριος με έχει το λόγο. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Ο πρόεδρος ε, μας έδωσε μια ενδελεχή και πολύ διαφωτιστική εικόνα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. For me, uh, Το ίδιο ισχύει και για μένα. Από κοινού συντάξαμε τη δήλωση αυτή. Μας κάλυψε πλήρως ο προλαλής σας. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Κατά τα άλλα, αυτά που μας παρουσιάζονται εδώ πέρα στο έγγραφο με τη θέση σας ε, αποτελούν λοιπόν αυτά μια πολύ καλή βάση για τις μελλοντικές εργασίες. Νομίζω ότι οι επιτροπές στις οποίες έχουν τα άτομα επαφής τους οι οργανισμοί θα πρέπει να μελετήσουν το έγγραφο αυτό τοποθέτησης και να τα λάβουν όλα αυτά υπόψη. Και να έχουμε πάντα φυσικά κατά νου τους οργανισμούς και τα περιστατική μας Επιτροπή. Μιλήσατε για τον οδικό χάρτη και για τις 90 δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πιο στενή συνεργασία και κατάρτιση προγράμματος ε, προγραμμάτων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν, αλλά θα σας λείπει ο διάλογος και η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπήρχαν, υπεγράφει η κοινή προσέγγιση από το Κοινοβούλιο και από, όλες, ε, τις, από όλους τους οργανισμούς, κατόπιν όμως ε, η σχετική ομάδα εργασίας εδώ στο Κοινοβούλιο διαλύθηκε. Νομίζω ότι η καλύτερη λύση θα ήταν να γράψετε μια επιστολή προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να παρουσιάσετε πώς έχει η κατάσταση και να δηλώσετε ότι το χρειαζόμαστε ένα όργανο επαφής στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό ο πρόεδρος θα το συζητήσει με τους πρόεδρους των ομάδων και θα βρεθεί μια λύση. Και τελικά θα αριστεί, πιστεύω, το αντίστοιχο όργανο επαφής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είπατε ότι δεν είσαστε ικανοποιημένοι με την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό του 2014 και ότι πιστεύετε ότι ελοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων των οργανισμών με τον προπολογισμό αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια πρόταση. Κοιτάξτε, να σας το πω ότι μπορεί να ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα αν δείτε τι συζητιέται αλλά και τι γράφεται στο Συμβούλιο. Πώς ξανά και ξανά γίνεται απόπειρα να περικοπεί ο προπολογισμό των οργανισμών, ειλικρινά θα σα σηκωστεί η τρίχα όρθια. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό, κατεπηγόντως, κατεπηγόντως, δεν ξέρω πώς και με τη μορφή ακριβώς, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι θα πρέπει να πάμε στα Υπουργικά Συμβούλια, στους Υπουργούς Οικονομικών Οικονομίας, προκειμένου τουλάχιστον να τους ενημερώσουμε να έχουν μια τοποθέτηση εδρωμένη, σωστά εδρεωμένη για το τι συζητείτε στην παρούσα φάση. Τι να σας πω, αυτά που πραγματικά ε, διαμείβονται τώρα είναι φρετά. Και θα ήθελα να πω ότι εν μέρει ευθύνεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι υπάλληλοι σε ό,τι αφορά δηλαδή την εντύπωση που επικρατεί στο Συμβούλιο για τους οργανισμούς. Γιατί, Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει ισολογισμούς που καταδεικνύουν ότι οι οργανισμοί σε αυτή την χρηματοδοτική περίοδο παίρνουν συν 4% σε σχέση με την προηγούμενη. Μα από ιστορική άποψη μπορούμε να μιλήσουμε για πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Το, πριν από χρόνια είχαμε 9 οργανισμούς. Τώρα έχουμε, το 2012 έχουμε 29, τώρα έχουμε 33 οργανισμούς. Ε, σας παρακαλώ. Και ξέρετε, αυτά δεν πέφτουν από τον ουρανό. Αυτό το κείμενο έχει συζητηθεί τόσες πολλές φορές. Αυτή η φράση, ότι αυτά δεν πέφτουν από τον ουρανό, οι υφιστάμενοι οργανισμοί έχουν όλοι μια νομική βάση. Αυτή η νομική βάση έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μάλιστα σε ορισμένε περιπτώσει ούτε καν μετά από πίεση του νομοθέτη. Τι έχει εφεύρει σε πολλέ περιπτώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σα πω ότι τη Δευτέρα το βράδυ μίλησα με κάποιον από τη Γενική Διευθύνση Περιβάλλοντος και ζητά κατεπηγόντως έναν οργανισμό για την περιβαλλοντική νομοθεσία και τον έλεγχο της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μιλάμε δηλαδή για άλλον οργανισμό. Κανείς από τους συναντέλφους δεν είναι κατά της δημιουργίας ενός τέτοιου οργανισμού και της έντρασης αυτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όντω δεν μπορεί να ελέγξει με συνέπεια την εφαρμογή τη σχετική νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα παράδειγμα σα δίνω. Παρ' όλα αυτά, στο Συμβούλιο τι λέει. Α, κοιτάξτε, αφού όλοι κάνουν περικοπέ, να κάνουν περικοπέ και οι οργανισμοί. Και τελικά, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενισχύει αυτή την τάση για εξωτερική διαμορφώση και ανάθεση όλων αυτών των ζητημάτων. Δεν ξέρω πόσο καιρό, πόσα χρόνια είμαι υπεύθυνη για τους οργανισμούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει και αναθέτει εξωτερικά τις αρμοδιότητές της και φυσικά αυξάνονται και οι αρμοδιότητες στα πλαίσια της κατηγορίας 5 μας μιλούν για εκτελεστικούς οργανισμούς, μας εξηγούν γιατί λειτουργούν καλύτερα έτσι τα πράγματα. Και όλα αυτά προκύπτουν και από τον ε, προϋπολογισμό των εφαρμοστικό και μετά υπάρχουν και οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί οι οποίοι φορτώνονται διαρκώ με νέε αρμοδιότητες, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και πολλές φορές με άλλες ε, διαδικασίες, με νομοθεσία την οποία εμείς εδώ αποφασίζουμε. Αλλά παράλληλα πρέπει να μην αυξηθεί το προσωπικό τους, να περιοριστούν τα κονδύλια τους, μα πώς θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό ότι δεν είναι δυνατόν. Είναι πραγματικά παράνοια αυτό. Και τώρα το λόγο έχει ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον Μασίλ για την παρουσίασή του. Εστενίζομαι πλήρως στα σχόλια της Γιούτα. Δεν έχω να προσθέσω ούτε να αφαιρέσω τίποτα. Οι ευρωβουλευτές, ιδιαίτερα στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, μεριμνούν ιδιαίτερως για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα έχουν επίγνωση των περιορισμών που υπάρχουν. Αλλά ως Ευρωβουλευτές συμβάλλουμε με το έργο μας στις Επιτροπές στην οικοδόμηση της Ευρώπης με διάφορα κείμενα προκειμένου να ενισχύσουμε την ολοκλήρωση, την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, τις ικανότητες και σε αυτό το κείμενο πολλές ε, ε, σε αυτή την προσπάθεια πολλές τις αρμοδιότητες αναθέτουμε στους οργανισμούς. Και θα αναφερθώ σε δύο παραδείγματα χαρακτηριστικά. Καταρχήν, ε, οργανισμός για την ασφάλεια της εναέρειας κυκλοφορίας. Ουσιαστικά αυτό χρηματοδοτείται ο οργανισμός αυτός. Εξασφαλίζει πιστοποίηση των επιχειρήσεων και από εκεί αντλεί τους πόρους του. Η πρόταση ε, που κάνουμε στον οργανισμό αυτό είναι να καταργήσει φέτος 10 θέσεις και μέχρι το 2017 να καταργήσει 50 θέσεις. Μιλάμε για θέσεις εμπειρογνωμόνων και ουσιαστικά οι εμπειρογνώμονες αυτοί πιστοποιούν ε, τις ε, εταιρείε και έτσι συμβάλλουν στην χρηματοδότηση του οργανισμού. Οπότε με την κατάργηση των θέσεων εργασίας στον οργανισμό θα μειωθούν οι πόροι, άρα θα χρειαστεί να αναθέσει σε εξωτερικούς ε, παράγοντες το έργο της, κάτι που θα αυξήσει το κόστος και για τους ε, φορείς της ενέργειας κυκλοφορίας και για τις ε, αεροπορικές εταιρείες, θα μειωθεί η ανταγωνιστικότητά τους και μάλιστα μια στιγμή που ο κλάδος αυτός βρίσκεται σε πλήρη άνθηση. Ενώ οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προβλήματα αναδιάρθρωσης και χαμηλής ανταγωνιστικότητας απέναντι στις εξωκοινωτικές εταιρείες. Οπότε όχι μόνο δεν κάνουμε οικονομίες με τις στάσεις αυτές και καμία προσπάθεια ολοκλήρωση, αλλά ταυτόχρονα στα κράτη-μέλη, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν έχουμε πια δυνατότητα καν Οπότε το μέτρο αυτό που είναι οριζόντιο για απολύσεις στον οργανισμό, μειώνονται οι πόροι του οργανισμού, μειώνεται η εμπειρογνωμοσύνη του και μάλιστα δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς γιατί δεν έχουν τα κράτη-μέλη τέτοια εμπειρογνωμοσύνη. Θα μειωθεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου των μεταφορών. Εξηγήστε μου λοιπόν πού έγκυται το πλεονέκτημα αυτή τη σύσταση. Είναι ανόητη από κάθε άποψη και από δημοσιονομική και από την άποψη σε ενέργειε κυκλοφορίας αλλά και από οικονομική άποψη η σύσταση είναι ανόητη. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω το λόγο τη. Δεύτερο παράδειγμα. Ο Μαρσέλ Βερσλίπ, ο πρόεδρο. Ε, είναι πρόεδρος της, του οργανισμού για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και μάλιστα συνεχίζεται η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του τέταρτου σιδηροδρομικού πακέτου για τις σιδηροδρομικές μεταφορές που είναι το 10% ουσιαστικά του Ευρωπαϊκού ΕΠ και οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες αφορούν όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα και προτείνουμε ένα τεχνικό πυλώνα που θα μεταφέρει στον οργανισμό που αυτή τη στιγμή είναι οργανισμός ε, ε, προτυποποίησης, ε, εναρμόνιση μάλλον των προδιαγραφών, όλα τα θέματα της πιστοποίησης και διαλειτουργικότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αντάλλαγμα, τι πόρους προσφέρουμε. 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για δύο χρόνια γελίο ποσό, δεν αξίζει καν... 500.000 ε, ε, συγγνώμη ευρώ το χρόνο, δηλαδή ε, γελίο ποσό δεν, δεν αξίζει καν να το συζητούμε. Ενώ αυξάνονται κατακόρυφα οι αρμοδιότητες του οργανισμού, το φόρτο εργασίας και η ευθύνη του οργανισμού. Οπότε προτείνουμε 20% αύξηση του, δυνα... του του προσωπικού μέσα σε πέντε χρόνια. Αλλιώς δεν θα εξασφαλίσουμε καμία διαλειτουργικότητα και βελτίωση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Και το νομοθετικό έργο του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στηρίζονται σε μια ουτοπική πραγματικότητα σε ό,τι αφορά το έργο αυτού του οργανισμού. Δεν θα καταφέρει καθόλου να ανταπεξέλθει στο, στο έργο. Και σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές έχουμε 150 υπαλλήλους ε, στον οργανισμό αυτό που κάνουν τεράστιο έργο ολοκλήρωση ε, και προτυποποίηση. Τώρα, με την αύξηση των αρμοδιοτήτων και την διάβηση και στην πιστοποίηση προτείνεται αύξηση του προσωπικού κατά 40 υπαλλήλους. Ελάχιστη αύξηση λοιπόν. Διαφωνώ με την πρόταση είναι παράλογοι, οικονομικά πρόσφοροι, ως προς την ασφάλεια κατάλληλοι και ανόητοι σε όλα τα επίπεδα. Τώρα δεν ξέρω αν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να καφιέται για υποτιθέμενες ε, επιτυχίες νομοθετικές που καταλήγουν όμως ε, σε ε, ανέφικτες συστάσεις. Πολλαπλασιάζουμε την έγκριση μέτρων, διατάξεων, οδηγιών και κανονισμών που όμως δεν έχουν αντίκρισμα στην πραγματικότητα. Και πολύ σωστά είπε η Πρόεδρος ότι το, το πρόβλημα των οργανισμών θα πρέπει να έρθει στο προσκήνιο των συζητήσεων γιατί διακυβεύει την αξιοπιστία των εργασιών μας και της Ένωσης. Αλλιώς θα συνεχίζουμε την ε, θέσπιση κειμένων που είναι ανέφικτα στην εφαρμογή. Το θέμα των οργανισμών, επαναλαμβάνω, έχει κεντρικό ρόλο και για τα θεσμικά όργανα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά ήταν δύο πολύ καλά παραδείγματα τα οποία γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, Ντομινίκ. Υπάρχουν πολλά περισσότερα παραδείγματα. Αλλά όπως σας είπαμε έχουμε και, άλλα, και άλλους οργανισμούς. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τους εκπροσώπους για την έκθεση, την, τις εκθέσεις τους. Σκούρα τα πράγματα. Πάντως, το πρώτο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι οι βασικές δαπάνες των υπηρεσιών είναι λειτουργικές, ε, επιχειρησιακές, όχι διοικητικές. Δεν πρέπει λοιπόν να εκτίθενται την σε περικοπές που σχετίζονται με τις διοικητικές διαδικασίες. Είχαμε μια σειρά παραδειγμάτων. Αν θέλεις να κάνεις εξοικονομήσεις στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να γίνει με αξιολόγηση. Προφανώς αξιολογούνται πάντα οι δομές και κάνεις μια σειρά διαθώτικών αποφάσεων. Άλλοι ας πούμε συζητούν να φύγει το ΣΥΠΟΛ από την Βρετανία και να πάει. Αλλά και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο αντιτίθεται ο κόσμος. Εδώ έχεις περιπτώσεις δηλαδή όπου μπορεί να έχεις εξοικονομήσεις, εν τέλει όμως κανείς δεν το θέλει. Και άλλες περιπτώσεις υπάρχουν όταν, ε, όπου συγχωνεύοντας κάποιες υπηρεσίες μπορείς να βελτιώσεις την αποτελεσματικότητα. Αλλά αυτό είναι δύσκολο όταν όλο αυτό σχετίζεται με την πολιτική κατανομή. Δηλαδή ένα, ένας αρχηγός κυβέρνησης θεωρείται ότι επιτυγχάνει όταν ε, ε, παίρνει μια υπηρεσία στη χώρα του. Αυτό δεν μπορεί να το αφήσει. Επίσης, σωστά τονίσατε ότι η Επιτροπή έχει μια λογική πρόταση Εμείς μπορούμε να πούμε ότι δεν μας ικανοποιεί η πρόταση της Επιτροπής, αλλά το Συμβούλιο κάνει οριζόντιες περικοπές και αυτό μπορεί να αντιμετωπίσουμε τώρα και νομίζω ότι η συζήτηση θα είναι δύσκολη. Μία ερώτηση έχω. Συχνά βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα σε κάποιες υπηρεσίες γιατί δεν έχουν οργανογράμματα. Ή γιατί δεν έχουν εφαρμοστεί τα οργανογράμματα. Κάτι που περιγράφηκε είναι ότι κάποιες υπηρεσίε έχουν τόσο μεγάλη περικοπή που δεν μπορούν να καλύψουν τα οργανογραμματά τους. Και εδώ θα ήταν χρήσιμο να έχουμε πληροφορίες γιατί είναι σημαντικό εν τέλει. Προφανώ θα πρέπει τι επόμενε μέρε να έχουμε μια σωστότερη εικόνα τη κατάσταση των αναγκών. Ξέρετε ότι το πρόβλημα των υπηρεσιών ήταν έλλειψη ενδιαφέροντος και κατανόησης του τι κάνανε. Αλλά όλο και περισσότερο οι εξειδικευμένε επιτροπές καταλαβαίνουν ποια είναι η κατάσταση και θα έπρεπε να στηριχθούμε σε αυτές για να μας βοηθήσουν με τις πληροφορίες τους. Εν γέννη, πάντως η εικόνα που έχω είναι ότι στο Συμβούλιο δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες. Το είδαμε όταν συζητούσαμε την κοινή συνεννόηση. Δύσκολο μπορούσε να βγει εντολή από το Συμβούλιο, διότι δεν ήξεραν τι έπρεπε να σκεφτούν για τα θέματα αυτά. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα. Σίγουρα είναι λάθος να βάζουμε όλες τις υπηρεσίες κάτω από το ίδιο καπέλο. Είναι τελείως τυχάρπαστο. Υπάρχουν υπηρεσίε και υπηρεσίε. Υπάρχουν νέε υπηρεσίε στον τομέα τη χρηματοοικονομική εποπτεία που έχουν τεράστια προτεραιότητα και είναι δύσκολο να ξεκινάς κάτι και μόλις ξεκινάει να του κόβεις τα φτερά. Η ειδική κατάσταση έχει να κάνει με τις υπηρεσίες που πληρώνονται με κατάθεση αιτήσεων ας πούμε που βγάζουν λεφτά δεν μπορεί να κάνει εκεί περικοπέ. Αυτό είναι περίεργο. Το κοινοβούλιο, μπορώ να σα πω, είχε κάνει μια μελέτη για τα τέλη που έφεταν οι υπηρεσίε, για δύο υπηρεσίε μιλούσαμε τότε. Το OHEM που έχει πλήρη χρηματοδότηση και την υπηρεσία φαρμάκων που χρηματοδοτείται από εξωτερική πληρωμή εν μέρη. Εδώ έγινε μια Η τιμολογιακή πολιτική τους γίνεται με πολιτική απόφαση και είχαμε μια συζήτηση επί της αρχής για την τιμολογιακή πολιτική και τι θα γίνει με στο μέλλον αν έχουν πλεονάσματα, αν έχουν ελλείμματα για να εξασφαλίζουμε ότι μπορούν να πληρώνουν τα κριτήρια που τους έχουν τεθεί. Διότι εγώ με την κατάσταση τώρα προβλέπω ότι όλο και περισσότερες υπηρεσίες θα χρηματοδοτούνται μέσω τελών ή προμηθειών στο μέλλον, όπως στον τομέα του χρηματο... της χρηματοοικονομικής εποπτείας. Ίσως το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο να μπορέσει να μπει στη μέση διάταξη της Επιτροπής και να γίνει μια γενικότερη συζήτηση για την έκθεση, ούτως ώστε να τεθεί και το θέμα των αρχών που θα τίθενται για την επιβολή ε, τελών. Σας ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει είναι. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα λίγο να αντιταχθώ, να μην εκνευριζόμαστε τώρα για θέματα τα οποία ακόμα δεν έχουμε καμία πρόταση μπροστά μας. Δύο ερωτήσει να κάνω. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις ε, της αλλαγής του κανονισμού για το προσωπικό για τους οργανισμούς, σε ό,τι αφορά τον ορισμό των 40 ωρών εβδομάδα, ε, Και παραλλήλου μιλάμε για αύξηση του προσωπικού. Η αλλαγή του κανονισμού λοιπόν πώς θα επηρεάσει του οργανισμούς. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Μια άλλη τώρα ερώτηση. Στην παρούσα φάση εξετάζουμε και τον προπολογισμό για τις ε, οργανισμούς και με εκπλήσει το πόσο περιορισμένο είναι το input. Πόσο συμμετείχαν λοιπόν ε, τα ίδιοι οργανισμοί για τον κανονισμό την αλλαγή του κανονισμού και την αναθεώρηση. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε. Γιούτα, κάτι άλλο. Ήμουν μέλλον της ομάδας εργασίας και αυτά που λες ε, πραγματικά με βρίσκουν σε μεγάλο βαθμό σύμφωνη Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να σκεφτεί πώς θέλει να τοποθετηθεί σε αυτό το μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό τοπίο. Αν ε, θέλουν όλο να απελευθερώνουν το δικό τους χρόνο και να έχουν όλο και πιο πολύ ελεύθερο χρόνο να το κάνουν. Αλλά σε τελική ανάλυση γιατί τους χρειαζόμαστε. Θα πρέπει σίγουρα να περιορίσουμε το εύρος των οργανισμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλαμβάνει τα νέα της καθηκόντα θα πρέπει να ακολουθούμε πολύ πιο πολυπρεριστική γραμμή σε ίδρυση νέων οργανισμών από ό,τι κάναμε ως τώρα. Ίσως θα έπρεπε να αναγκάσουμε το Συμβούλιο να κάτσει να ανοίξει όλες τις νομικές βάσεις για τους οργανισμούς και θα ήθελα να συμβεί αυτό. Αυτό για το άνοιγμα της νομικής βάσης, για την καλύτερη εξοπλισμό και χρηματοδότηση των οργανισμών, γιατί σίγουρα κάθε οργανισμός έχει διαφορετικά προβλήματα. Θα πρέπει πραγματικά να κάτσουμε να εξετάσουμε τη νομική βάση εκ νέου και ως Επιτροπή Προπολογισμών θα πρέπει να το προβάλλουμε αυτό και μάλιστα με στεναρότητα προς, τους, προς το Συμβούλιο για να βοηθήσουμε τους οργανισμούς να βγουν από αυτό το τέλμα των προβλημάτων που τους μαστίζουν και που δεν αλλάζουν και ποτέ. Σπάνια στη ζωή μου έχω λάβει τόσο σωστές και ακριβείς πληροφορίες όσο από την διαθεσμική ομάδα αυτή για τις ε, οργανισμούς. Όλα τα στοιχεία που διάβασα στο έγγραφο τοποθέτηση ήταν πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμα. Μα ξέρουμε τι χρειάζονται οι οργανισμοί. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να του βοηθήσουμε. Α το κάνουμε επιτέλου. Είναι, λέει η πρόεδρο, κάποια από τα καλά μας ε, σχέδια πολύ απλά δεν πέρασαν στο Συμβούλιο. Αυτό είναι σαφές. Η Μόνικα έχει το λόγο. Καταρχάς θα ήθελα να συμφωνήσω με την κυρία Γέντσεν. Όντως, η επιμονή του Συμβουλίου και των κρατών μελών όταν έχει δημιουργηθεί ένας οργανισμός να μην αλλάξει τίποτα. Είναι πραγματικά κάτι το απίστευτο κοιτώντα το θέμα του ΣΕΠΟΛ. Δεν επρόκειτο για μια πρωτοβουλία, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τώρα η Μεγάλη Βρετανία είναι αυτή που α, παρουσιάζει τα προβλήματα. Θα μπορούσαμε να, έχουμε, να το έχουμε σκεφτεί και από πριν για το πώς ε, μπορούν να συνδεθούν τα θέματα της Europol, της Eurojust, του Frontex πώς μπορούν όλα αυτά τα προβλήματα και τα θέματα να συνδεθούν. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κάνει αυτό μόνο όταν έρθει συνήθως ένα κράτος μέλος και πει ότι δεν θέλει πλέον να συνεχιστεί η κατάσταση και τότε ξεκινάνε τεράστιες συζητήσει. Γιατί τελικά τα στυλώνουν οι Βρετανοί και λένε ότι τελείω θέλουμε να πουλήσουμε το κτίριο, δεν έχουμε χώρο για σας πλέον και δημιουργούν προβλήματα. Αυτό θα έπρεπε να έχουμε κάτι να το σκεφτούμε πολύ πιο νωρί για θέματα δικαιωμάτων ε, των γυναικών, των ανθρώπων. Κατά πόσον έχει νόημα να συνδέονται αυτά τα δύο θέματα. Θεωρώ ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τα δικαιώματα των ανθρώπων. Και θεωρώ λοιπόν ότι εν μέρει οι δύο οργανισμοί κάνουν το ίδιο έργο. Επικαλύπτονται οι τομεί αρμοδιότητας με κάποιες φυσικά αποχρώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τι βαθμό ε, έχει πάρα πολύ δίκιο είναι που το ρωτάει. Σε ποιο βαθμό λοιπόν ορίζει τον ίδιο της το ρόλο και πώς τον ορίζει το ρόλο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να αναφερθώ σε έναν οργανισμό και να μην πω ποιο, ποια γενική ε, διεύθυνση μου το είπε αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά λίγο πολύ μου είπε η Γενική Διεύθυνση ότι ο οργανισμός είναι πιο μεγάλος από την Γενική Διεύθυνση. Αυτό σε επίπεδο εθνικού κράτους μέλους είναι λογικό. Ε, το οργανωτικό κομμάτι είναι πιο μικρό από το εκτελεστικό. Αυτό έλειπε να είναι πιο μεγάλα τα υπουργεία από τους αντίστοιχους εκτελεστικούς οργανισμούς. Όντως λοιπόν, έχω το εξή πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ορίζει με ακρίβεια και σαφήνεια ποιες ε, αρμοδιότητες εκτελεστικές αναθέτει στους εξωτερικούς οργανισμούς. Τα θέματα Europol δεν μπορεί να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλάμε για συντονισμό αστυνομικών δυνάμεων. Δεν είναι αυτό καθήκον της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σαφέ. Αυτό πραγματικά χρειάζεται να το κάνει ένα εξωτερικό οργανισμό. Υπάρχουν όμως ε, οργανισμοί οι οποίοι θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερα εξοπλισμένοι, να έχουν για παράδειγμα πιο καλή χρηματοδότηση. Όταν μιλάμε ε, για οργανισμό καταπολέμησης της ε, φοροδιαφυγής, και δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό γιατί, για παράδειγμα, είναι μόνο 12 τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τον συντονισμό 27 κρατών μελών. Προφανώς τα προβλήματα όπως η φοροδιαφυγή θα συνεχιστούν. Και σας το λέω αυτό ότι μόνο 10% να γλιτώναμε από την φοροδιαφυγή θα μπορούσαμε να προσλάβουμε δεν ξέρω και εγώ πόσους ε, επιπλέον εργαζόμενους ε, και έχει απόλυτο δίκιο η Αν Γένσεν. Κοιτάξτε, για παράδειγμα τώρα δημιουργούμε ένα κέντρο για την καταπολέμηση του εγκλήματος και η Europol έχει εννέα άτομα λιγότερα. Ε, εντάξει, τι να σας πω, καλή επιτυχία. Θα χαρούν μια χαρά οι εγκληματίες, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει κανένας να τα καταπολεμήσει όλα αυτά. Τρία άτομα έχουμε μόνο για την καταπολέμηση της παιδικής προγραμματίας στο διαδίκτυο. Συγχαρητήρια Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν τα καταγγείλουμε αυτά, τι μας λένε, ότι Α, κοιτάξτε, η Γυροπόλα έχει πάρα πολύ προσωπικό. Μα δυστυχώ τόσο ευρύ είναι το φάσμα των εγκλημάτων. Χρειάζεται συντονισμό. Χρειάζονται άτομα. Αυτό δεν αφορά μόνο τη Γυροπόλα αφορά και πάρα πολλού άλλου οργανισμού. Τη Eurojust, παράδειγμα συντονισμό των δικαστικών αρχών. Κάτι πρέπει λοιπόν να γίνει στα πλαίσια της Eurojust. Δεν είναι δυνατόν να τρέχουν όλα αυτά χωρίς χρηματοδότηση. Σωστό και το ερώτημα με τις 40 ώρες την εβδομάδα. Αυτό είναι κάτι αναπόφευκτο. Αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να διαχωριστεί από τον τομέα των νέων αρμοδιοτήτων και θα πρέπει να πω να πω το εξή. Όταν χρειαζόμαστε ένα οικοδόμημα όπως το ICC, θα πρέπει να οριστούν όλα αυτά εκ νέου. Και να υποδηλώσουμε ότι πρόκειται για έναν οργανισμό σε ανάπτυξη. Και αυτό από τώρα θα πρέπει να το πούμε. Ο τρόπος επίσης ορισμού της ανάπτυξης ενός οργανισμού και αυτός είναι πολλές φορές ε, παράλογος. σαφές το θέμα. Με τις 40 ώρες θα πρέπει να το υπολογίσουμε επακριβώς. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να εξετάσουμε ποιες αρμοδιότητες θέλει να ε, διατηρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα τέλη για την καταχώρηση σε έναν τομέα μιας μικρής επιχείρησης, επιβάλλονται σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι και 9.000 ευρώ Και όσο πιο, πολλές, πιο πολλά είναι τα τέλη, όσο πιο υψηλά είναι τα τέλη, τόσο πιο καλά δημιουργεί ένας οργανώσεις, ε, οι οργανισμοί. Αλλά κανείς φαίνεται να μην ε, ενίσταται και να ε, λέει ότι αυτό επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις οποίες προσπαθούμε να υποστηρίξουμε. Μία τέτοια ανάλυση λοιπόν θα την ήθελα κατεπηγόντως και θεωρώ ότι πολλές από τις δράσεις μας είναι κατακαιρματισμένε και αντιφαντικές. Και τώρα που είναι εδώ η Τρόικα, τουλάχιστον να λάβουμε κάποιες επιπρόσθετες υποδείξεις από πλευρά σας ό,τι αφορά τέτοια θέματα προϋπολογισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Γιούτα Χάουκ. Αλλά αυτό που λες ότι όσο πιο πολλά είναι τα τέλη, τόσο καλύτερα λειτουργεί ο οργανισμός, μα αυτό από μόνο του είναι παράλογο, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει ακόμα και στον τομέα που χρηματοδοτείται από τα τέλη να, περικο... να κάνει περικοπές. Δηλαδή, ο κλάδος, η βιομηχανία θέλει να γίνεται σωστή δουλειά. Θέλει να πληρώνει. Αλλά όταν δεν υπάρχει κόσμος, αν δεν υπάρχει προσωπικό, γιατί μέσω του offsetting αφαιρούνται ακόμα και άτομα από την αίμα που χρηματοδοτείται από τα τέλη και δεν μπορούν τελικά να έχουν τις υπηρεσίες αυτές. Ποιος πρέπει τελικά η καινοτομία. Μία μικρή παρατήρηση. Η κυρία Χόλμαϊρ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παρέχει σε αυτή τη φάση μόνο contract agents, συμβασιούχους, οι οποίοι δεν μπορούν, για παράδειγμα, να περιλαμβάνουν ε, εμπειρογνώμονε από τα κράτη-μέλη. Γιατί ποιος θα έρθει ε, για 3.000 ευρώ το μήνα να έρθει να κάνει για κάποια χρόνια αυτή τη δουλειά. Δεν μπορούμε λοιπόν ούτε temporary agents, ούτε ε, προσωρινούς συμβασιούχους να προσλάβουμε. Όλα θέλει να τα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με contract agents. Ναι, ναι, ναι, αυτά είναι πάρα πολύ ενσυχητικά, λέει η Πρόεδρο Γιώτα Χάουγκ. Η δική μου ερώτηση είναι κατά πόσον η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνάδει με τους κανόνες με τους οποίους ε, και είναι συμβατή με τους κανόνες με τους οποίους ε, καταρτίζεται ο προπολογισμό. ή μήπως είναι και παράνομη, αντίθετη στον νόμο ναι, ναι, ναι, σας παρακαλώ να μας απαντήσει, κύριε Σπιέτσα. Αν ε, μέσα από όλες τις κατηγορίες κοιτάξω τις ε, οργανισμούς και πω ότι ωραία, αυτοί είναι οι οργανισμοί μου τόσο προσωπικό που ασχολούν. Και 1% θα πρέπει, κατά 1% να, πρέπει να μειώσουν το προσωπικό και το 1% του προσωπικού τους πρέπει να το αναθέσουν σε ένα πουλ προσωπικού και από αυτό το πουλ και από αυτό τον λοιπόν οργανισμοί άλλης κατηγορίες ε, οι οποίοι δημιουργήθηκαν σε άλλη φάση και προβλέπεται να επεκταθούν, εμπασχετώσει που πρέπει να έχουν περισσότερο προσωπικό, ε, μπορούν να πάρουν για παράδειγμα άτομα από την κατηγορία 1α για να τους στείλω στην κατηγορία 3, είναι δυνατόν. Δεν είναι αυτό καν αντίθετο στον νόμο, εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε χρήματα σε μία κατηγορία να τα μεταφέρουμε έτσι απλά σε μία άλλη κατηγορία, όποτε θέλουμε. Το ερώτημα της είναι Γκρέσλε. Εγώ δεν μπορώ να το απαντήσω. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, έπρεπε να την απαντήσει. Ε, αν θέλετε να την απαντήσετε, πείτε μας για την αλλαγή του κανονισμού, την τροποποίηση του κανονισμού, πώς θα επιδράσει και πώς θα επηρεάσει α, με τους οργανισμούς και τι γίνεται και με την αλλαγή στον προπολογισμό, με, με την διαμόρφωση του προπολογισμού. Uh, Ευχαριστώ. πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρώτη σας ε, σύσταση, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε συνομιλητή του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα στείλουμε σχετική επιστολή στον Πρόεδρο Σούλτς. Είπατε ότι τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο επιμένουν για περαιτέρω μείωση του προϋπολογισμού των οργανισμών σας διαβεβαιώ ότι στο δικό μας επίπεδο και να δώσω ε, το λόγο και στους συναδέλφους που προσπάθησαν με κάθε τρόπο να σε εξηγήσουν γιατί όχι μόνο δεν θέλουμε μείωση, αλλά ζητούμε και διεύρυνση και είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η μείωση. Και να σας δώσω ένα απλούστο παράδειγμα. Αναφέρθηκε ο Οργανισμός για τους Σιδηροδρόμους σε λίγο χρόνια θα αναλάβουμε και το θέμα της έγκρισης ε, και του τροχαίου υλικού σιδηροδρόμων στην Ευρώπη. Και τα κράτη-μέλη έχουν περιορίσει τις αρμόδιες αρχές ε, ε, και τους περιπολογισμούς τους σχετικά. Κύριε Ρικέ, τα επιχειρήματα και τα παραδείγματα που μας παρουσιάσατε είναι πάρα πολύ εύστοχα και εύγλωτα. Αναφέρθηκαν πολλές δυσκολίες και από άλλους ευρωβουλευτές. Το θέμα είναι όταν ένας οργανισμός έχει, χρειάζεται περισσότερους υπαλλήλους και για να ανταπεξέλθει στο έργο της, δεν μπορεί πολλές φορές εξαιτίας τον περιορισμό να το κάνει. Και στα πλαίσια της, ε, των προσαρμογών εφαρμόζουμε μια επικίνδυνη πολιτική. Για παράδειγμα, ο κλάδος μας ζητά χρηματοδότηση για να διευρυνθεί ο οργανισμός και αυτό το θεωρεί απαραίτητο και ο κλάδος, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ούτε πόρους ούτε μέσα για να το κάνουμε. Επιπλέον, αναφερθήκατε κι εσείς και άλλοι ευρωβουλευτές στο γεγονό ότι σήμερα μας προτείνουν να χρησιμοποιήσουμε ε, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες, ενώ παράλληλα με την εφαρμογή της πολιτικής για την καταπολέμηση της σύγκρουσης συμφερόντων δεν μπορούμε να προσλάβουμε ε, εθνικούς εμπειρογνώμονες για να ε, διαθετήσουν διαφορές σε περίπτωση επιστοποίηση έγκρισης οχημάτων. Ούτε οι συμβασιούχοι είναι λύση παράδειγμα τι γίνεται με τους μηχανικούς που έχουν ε, δεκαετή, δεκαπενταετή διεθνή πείρα, μιλούν τρεις γλώσσες και χρειάζεται να περάσουν ε, τριετή έλεγχο για να δώσουν την έγκριση για ένα τρένο ε, μεγάλης ταχύτητας. Είναι δυνατόν συμβασιούχοι να μπορέσουν να αναλάβουν τέτοιες υπεύθυνε θέσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα τα διοικητικά έξοδα των οργανισμών, το είπε και δυστυχώς το επιβεβαιώνω, μας ενδιαφέρει ο στόχος της νέας προσέγγισης ε, για το δημοσιονομικό κανονισμό και τον κανονισμό του προσωπικού. Και είμαστε και εμείς υπέρ των στεύσεων ε, της απλοποίησης των κανόνων για τους οργανισμούς, γιατί ξέρετε ότι εμείς ε, πληρούμε όλους τους κανόνες που ισχύουν για τα υπόλοιπα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Και είναι πολύ δύσκολο, ειδικά για, τις, για, τους, για τους μικρούς οργανισμούς να τηρήσουν όλες αυτές τις διατάξεις. Σε ό,τι αφορά τη νέα πρόταση ε, του κανονισμού προσωπικού για την αύξηση των ωρών σε 40 εβδομαδιαίως. Δυστυχώς δεν συμμετείχαμε στις διαβουλεύσεις για τη μεταρρύθμιση του, του κανονισμού προσωπικού. Ε, βέβαια, <laughs> για τους 40 ώρες, μακάρι να δουλεύαμε μόνο 40 ώρες την εβδομάδα. Και αυτό ισχύει για όλο το προσωπικό. Σας διαβεβαιώ ότι ήδη το προσωπικό μας δουλεύει πολύ περισσότερο από 40 ώρες τη εβδομάδα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες παρατηρήσεις, συμφωνώ. Αλλά να δώσω το λόγο στον Μόρτον, γιατί νομίζω ότι έχει κάποια πιο γενικά σχόλια. Ευχαριστώ. Δύο σύντομες παρατηρήσεις Καταρχήν, ε, ποιος είναι ο ρόλος και η θέση των οργανισμών στην οικογένεια των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Θα πρέπει να γίνει σημαντική πρόοδος ε, στο να γίνει αντιληπτός ο ρόλος και η θέση αυτών των οργανισμών, γιατί δεν υπάρχει μια αντίληψη ε, για το ρόλο των οργανισμών και τη συμβολή τους στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να βελτιωθεί στη συζήτηση. Να δοθεί ο σωστός ρόλος και στη θέση στις ε, στους οργανισμούς. Γιατί μερικές φορές ακόμη και αρμόδιες αρχές στα κράτη-μέλη δεν ε, είναι εξοικειωμένε με το ρόλο των οργανισμών. ενώ οι περισσότεροι οργανισμοί βρίσκονται σε πρωτεύουσες κρατών μελών. Αυτό το συζητούμε στην Τρόικα. Πώς θα γίνει καλύτερη ενημέρωση ε, για τους οργανισμούς ώστε να υπάρχει κοινή ενιαία αντίληψη. Τώρα, αναφέρθηκε ένα σχόλιο για τη συνεργασία ε, των οργανισμών ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ε, ισότητας των φύλων. Αρχική απόφαση μιλούσε για δύο διαφορετικούς οργανισμούς. Πάντως υπάρχει μεγάλη συνεργασία και σε διοικητικό επίπεδο, θέματα διαγωνισμών, αλλά και σε ουσιαστικό επίπεδο. Οπότε αποφεύγουμε πάση θυσία επικάλυψη των προσπαθειών οι αντιφατικές ενέργειες. Αντίθετα έχουμε πολύ στενή συνεργασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι. Επειδή χρειαζόμαστε και την απάντηση του κυρίου Πρέζα, αλλά και επειδή πρέπει να μιλήσει και ο Γιάννη Πράτης για, την, ε, για τον προπολογισμό, θα μπορούσατε ίσως ε, να θέσετε τα ερωτήματά σας κατηδίαν. Μιλήσατε για 40 ώρες εργασίας και για το flex time που ακολουθούν οι οργανισμοί. Ποια είναι, ποιος είναι ο υπολογισμός, θέλω πιο συγκεκριμένα στοιχεία σας, παρακαλώ συγκεκριμενοποιήστε λίγο την απάντησή σας, δεν μπορώ με δύο προτάσεις να τα δεχτώ αυτά. Ο κύριος Πρίζα. Uh, Ευχαριστώ. Δεν θέλω να απαντήσω για την ευελιξία, για το flexi time. Ο συνάδελφος θα το απαντήσει. Για να επανέλθω στο πλαίσιο της πρότασης για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2014 και το πώς διαμόρφωσε την πρόταση αυτή η Επιτροπή. Στο σημείο 23 της Διοργανικής Συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία όπως έχει και επί της οποίας υπάρχει συμφωνία μεταξύ των τριών οργάνων αναφέρεται ότι οι διάφοροι θεσμοί και υπηρεσίε θα πρέπει να μειώσουν 5% της δαπάνης τα επόμενα 5 χρόνια. Το ίδιο φορά στην αύξηση στις ώρες εργασίας σε 40 ώρες την εβδομάδα. Η Επιτροπή διαμόρφωσε τις προτάσεις, τις προτάσεις της βάση των συμφωνιών για τα δύο δημοσιονομικά και δεν αρνούμε ότι υπάρχει μία ένταση μεταξύ των δημοσιονομικών διαδικασιών και υποχρεώσεων και των νομοθετικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Με αυτό το πλαίσιο είναι σαφές ότι η ύπαρξη υπηρεσιών σε διάφορα στάδια της ζωής τους, άλλες καινούργιες, άλλες παλιότερες, ενώ άλλες υπάρχουν μεν αλλά αυξήθηκαν οι αρμοδιότητές τους λόγω νομοθετικών αρμοδιοτήτων και αποφάσεων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, έχουν διαφορετικές ανάγκες. Αν θέλετε λοιπόν να αντιμετωπίσετε τις διαφορετικές αυτές ανάγκες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, με ένα μειούμενο πλαίσιο ανθρώπινου δυναμικού, Μπορείς να το κάνεις με γενική προσέγγιση. Αυτό έκανε και η Επιτροπή. Είδε τις διάφορες ε, καταστάσεις, εξέτασε ξεχωριστά το, τον κάθε οργανισμό, τον κάθε δομέα και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε στον προϋπολογισμό του 2014. Εφόσον δεχτείτε αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια στην πολιτική μας η Επιτροπή ακολουθεί τους προσανατολισμούς που περιλαμβάνει η Διοργανική Συμφωνία. Εκεί δεν υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ νέων δομών και υπηρεσιών ως προς την πήγη χρηματοδότησης. Ε, αναφέρεται σε, όλα τα, σε όλους φορείς και τις υπηρεσίες και υπάρχει ένα θέμα με ε, τις υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από ενωσιακή χρηματοδότηση αλλά η ίδια συλλογιστική μπορεί να γίνει και για ε, τα τέλη που πληρώνουν οι οικονομικοί φορείς, διότι τα τέλη είναι ένα κόστος στην οικονομική, στον οικονομικό φορέα που καλύπτει τις ανάγκες του φορέα. Άρα υπάρχει ένας βαθμός ανάγκης Υπάρχει ένα, μια, ένας βαθμός ανάγκης βελτίωσης αποτελεσματικότητας και για αυτοχρηματοδοτούμενους φορείς. Δόθηκαν παραδείγματα με αναφορές σε συγκεκριμένα συγκεκριμένες υπηρεσίες ε, των οποίων οι αρμοδιότητες αυξήθηκαν, δόθηκαν κάποια παραδείγματα για την περίπτωση της υπηρεσίας ασφάλειας της αεροπλοείας το 2013 υπήρξε αύξηση σε 16 θέσεις. Άρα οι, οι υποχρεώσεις, οι υποχρεώσεις της υπηρεσίας αυτής αναγνωρίστηκαν. Στον προγραμματισμό για το 2020 λήφθηκαν υπόψη οι νέες αρμοδιότητες και άλλων υπηρεσιών. ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των μελλοντικών αναγκών, η κυρία Γέντσεν και η κυρία Χολμάγερ αναφέρθηκαν στη δυνατότητα που δικαιολογείται και είναι χρήσιμη συγχωνεύσεων ΣΥΠΟΛ και Europol ή άλλες περιπτώσεις υπηρεσιών που έχουν συνάφεια στις δραστηριότητε τους. Οπότε εμείς ξαναπάμε στην ένταση μεταξύ, στην απόκληση μάλλον μεταξύ αποτελεσματικότητας και άλλων υποχρεώσεων που μπαίνουν στην νομοθετική διαδικασία. Νομίζω ότι έχουμε ένα συλλογική υποχρέωση να προσπαθήσουμε να φέρουμε μαζί αντιφατικές ρυθμίσεις. Να πω και κάτι ακόμα. Είπατε κι εσείς πρόεδρε ότι όντως αυξήθηκε ο ρυθμός των υπηρεσιών. 32 είναι πια. Ήταν πια το 2013. Από το 2000 η Ευρώπη οχταπλασίασε την συνεισφορά της σε ό,τι φορά τις δαπάνες και τετραπλασίασε τη συνεισφορά της ως προς προσωπικό. Τώρα να απαντήσω στην ερώτησή σας για τις μεταβιβάσεις, τις μεταφορές ατόμων μεταξύ κατηγοριών. Δεν υπάρχει μεταφορά αυτό που προτείνει η Επιτροπή με το 1% αναδίπλωσης είναι η μείωση αριθμού, του αριθμού των θέσεων στο πρόγραμμα εγκατάστασης, κάτι που γίνεται για κενές θέσεις μόνο. Δεν υπάρχει κίνηση λοιπόν ατόμων, αλλά προσαρμογή του πλαισίου. Ούτε οι πιστώσεις κινούνται, υπάρχουν ενδεικτικά μικρά ανώτατα πλαίσια σε κάθε υποκατηγορία. Μέσα στα πλαίσια των ανώτατων αυτών ορίων η χρησιμοδοτήση όλων των υπηρεσιών πρέπει να καλύπτεται. Θα προσέφετα ότι η Επιτροπή πρότεινε την δημιουργία ενός νέου οργάνου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, καθάρι, ε, εξυγίασης των τραπεζών που θα πρέπει να είναι αυτοχρηματοδοτούμενη υπηρεσία. Ε, προφανώς θα πρέπει να υπάρχουν κονδύλια που θα καλύπτουν άλλες ανάγκες που μπορεί να προκύξουν μεταξύ τώρα και του 2020. Αυτά είναι ο Λίγης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σημειώνουμε λοιπόν τις απαντήσεις αυτές. Δεν μπορώ να πω ότι μας ικανοποιούν απόλυτα. Σας ευχαριστώ όλους. Όχι, δεν πρόκειται να παρευθυνθώ ακόμα κι αν έτσι ακούγεται. Όχι, σε καμία περίπτωση να σας ευχαριστώ, να σας ευχαριστήσω που ήρθατε ε, και φυσικά και την Ρόικα που πήρε το λόγο και τους διευθυντές που ήρθαν εδώ για να ακούσουν και που σιώπησαν ενδεχομένω, αλλά κάθισαν και σκέφτηκαν αυτά που έπρεπε. Κατρίν, σε αγγίζουν ίσως ιδιαίτερα σε αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα πρέπει να προχωρήσουμε το πρόγραμμα της Επιτροπής Προπολογισμών, γιατί σήμερα το απόγευμα δεν θα έχουμε πλέον μαζί μας ε, τον εισηγητή μας. Θα πρέπει να φροντίσουμε τα θέματα του προϋπολογισμού 4 και 5. Τα σημεία 4 και 5. έχεις το λόγο. Ευχαριστώ Γιούτα μια σύντομη ανασκόπηση των πολλών διορθωτικών προπολογισμών που έχουμε, διότι εγώ θα ξεκινήσω από τον διορθωτικό 2, θα μιλήσω για τον 3, τον 4, τον 5 και για όλες τις τρευλώσεις που θα κληθούμε σήμερα το απόγευμα να ψηφίσουμε. Διορθωτικός προπολογισμός υπαριθμών 2. Όπως θυμάστε, αυτός έχει μια μακρά ιστορία κάναμε μια πολιτική, λάβαμε μια πολιτική απόφαση στις 7 Μαΐου, εγκρίνοντας δύο δόσεις, 7,3 δις η πρώτη και μια δεύτερη μετά την οποία θα έπρεπε να υπήρξε και ένας επιπρόσθετος διορθωτικός προϋπολογισμός. Στις 14 Μαΐου υπήρξε πολιτική συμφωνία για το, την πρώτη δόση του διορθωτικού προϋπολογισμού 2, ενώ μετά την έγκριση του δημοσιονομικού πλαισίου στις 9 Ιουλίου εγκρίθηκε η διανομή το 7,3 με διακατανομή των περικοπών σε όλες τις γραμμές αναλογικά που είχε προτείνει η Επιτροπή. Το Συμβούλιο δεσμεύθηκε επιπλέον να εξασφαλίσει την κάλυψη ενός περαιτέρου διορθωτικού προπολογισμού όταν εφόσον υπάρξει ανάγκη πληρωμών μέχρι τέλος του έτους. Πρόκειται για έναν προπολογισμό διορθωτικό που κατά την άποψή μου και το θεωρώ αυτό είναι αναγκαίο λόγω των αναγκών να υπάρξουν πλήρωμες για να κλείσει η χρήση 2013 και που από πλευράς μας ε, θα παραμείνει προϋπόθεση για να δώσουμε την υποστήριξή μας στο νομοθετικό πακέτο για το ΠΔΠ, το φθινόπωρο. Για τον διορθωτικό αυτό προπολογισμό είμαι υποχρεωμένο να αναφέρω στους συναδέλφους ότι η τροπολογία η προθεσμία υποβολή τροπολογιών είναι 16 Ιουλίου 12 το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε τον προπολογισμό 5 Σεπτεμβρίου και στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου κατόπιν. Παράλληλα με τον διορθωτικό τροποποιητικό προλογισμό υπαριθμών 2 έχουμε και τον υπαριθμό 3. Εδώ ο στόχος είναι αφορά το, πλεό, το ετήσιο πλεόνασμα που είναι 1,23 δις ευρώ και που επιστρέφεται, πρέπει να επιστρεφεί στα κρατημέλη μειώνοντας αναλογικά την συνεισφορά τους. Η έγκριση του προϋπολογισμού αυτού μειώνει προφανώς την εισφορά των κρατών μελών για την κάλυψη του διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμών 2, άρα το ποσό αυτό, ο προπολογισμό αυτό, θα πρέπει να σε αναφερθεί ως ε, δεόμενος πολιτικά με τον υπαριθμό 2. Προτείνω και εδώ να εγκρίνουμε τη θέση του Συμβουλίου της η Ιουλίου που επιβεβαίωσε την πρώτη της Επιτροπής χωρίς τροπολογίες. Και εδώ η προθεσμία για τις τροπολογίες προβλέπεται για τις 16 Ιουλίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Προπολογισμών 5 Σεπτεμβρίου και θα πάμε στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο πάλι. Κατόπιν, όπως έλεγε και η πρόεδρος Χάουγκ, έχουμε και τους διορθωτικούς τροποποιητικούς προϋπολογισμούς 4 και 5. Ο 4 αφορά μια πρόταση της Επιτροπής που θέλει να ενισχύσει τα οργανογράμματα των υπηρεσιών για το ευρωπαϊκό GNSS, την, ε, πλοή, την δορυφορική πλοήγηση δηλαδή, και την ΕΑΤΣΕΑ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Οπτικοκουσιών Μέτρων και το Δικαστήριο. Η, επιτροπή, η πρώτη επιτροπή είναι ουδέτερη για τον δημοσιονομικά, διότι η ενίσχυση των οργανικών θέσεων εκεί αντιστοιχίζονται με μηνύωση του προπολογισμού της Επιτροπής μέσα στους ε, πόρους που, είναι, που για το δικαστήριο. Για το GNSS, την υπηρεσία δορυφορικής πλοήγησης, υπήρξε έτοιμα 20 θέσεων ανάλογες με τις νέες αρμοδιότητες που έχει τον Καλλιλέο. Για το ΕΑΣΕΑ δε ζητούνται 15 ε, μόνιμες θέσεις και 2 έκτακτες θέσεις. Ενώ για το δικαστήριο το αίτημα είναι ένας γενικός εισαγγελέας και 7 μέλη προσωπικού του προσωπικού γραφείου. Για το δικαστήριο επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω και εξ του συναδέλφου Μπόρνα που λείπει σήμερα που είναι υπεύθυνο για, το, θέμα αυτό ότι δεν λήφθηκε υπόψη το αίτημα να υπάρξουν ε, προσλήψεις εννέα υπαλλήλων νομικών που θα μειώσουν την καθυστέρηση της εξέτασης των υποθέσεων. Αυτό δεν έγινε δεκτό από την Επιτροπή, ούτε αξιολογήθηκε και λήφθηκε υπόψη από υπολογισμό το 2014. Και εδώ προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 16 Ιουλίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει 5 Σεπτεμβρίου και η τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Διορθωτικός προϋπολογισμός 5 κάλυψη της εκμετάλλευσης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρώπης προς όφελος Κροατίας, Σλοβενίας και Αυστρία για 14,5 εκατομμύρια ευρώ. 14,6. Ο συνάδελφος κ. Φερνάντες σίγουρα θα προσθέσει κάποια ζητήματα για το θέμα αυτό, δεδομένου ότι αυτός παρακολουθεί την έκθεση. Ε, Παρότι επήγει το θέμα, και την πολιτική ψηφοφορία που λάβουμε... στις 27 Ιουνίου για να δείξουμε στο Συμβούλιο ότι είμαστε έτοιμοι να εγκρίνουμε αυτό το διορθωτικό προπολογισμό, το, Κονσίλιο, το Συμβούλιο συγγνώμη, δεν εξέφρασε την θέση του προς το παρόν. Έγκαιρα για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην Ολομέρεια του Ιουλίου. Θα ψηφίσουμε λοιπόν στις 5 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή Προπολογισμών και θα έχουμε την Ολομέλεια στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Και εδώ λοιπόν θα επικεντρώσουμε τις ψηφοφορίες μας τη συνάντηση Σεπτεμβρίου και κατόπιν στην Ολομέλεια. Αυτά ω προ τον, προς τους Αν θέλετε να μου δώσετε λίγο χρόνο να κάνω και λίγο σχόλια για τις επιστροφές. Όπως ξέρετε, οι ελλείψεις του προϋπολογισμού για τις πληρωμές, ιδίως δε η καθυστέρηση με τις οποίες εγκρίνει το διορθωτικό προπολογισμό παριθμών 2 θέτει σοβαρά προβλήματα στην Επιτροπή για την υλοποίηση κάποιων προγραμμάτων. Μας επιβάλλει λοιπόν να αξιολογήσουμε μια σειρά επιστροφών που προτείνει η Επιτροπή για να περάσει από τη γραμμή του προπολογισμού που υπάρχει κεφάλαιο σε εκείνες τις γραμμές όπου όχι μόνο δεν υπάρχει κάλυψη αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις τι συμβαίνει. Για κάποια από αυτά τα θέματα δε είμαστε υποχρεωμένοι να μιλήσουμε για τις καθυστερήσεις με τις οποίες εκφράζουμε, ε, ε εκφράζουμε τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ευρώπη. Θα μιλήσω ότι η μεταφορά 4 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση του προγράμματος ΙΖΑ διαλειτουργική λύση για την Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση στο 1α. Λόγω της έγκλησης των διορθωτικών προϋπολογισμών 2. Στον προϋπολογισμό του 13 η μείωση οδήγησε σε σε πλήρη έλλειψη πόρων. Επ' αυτού νομίζω ότι υπάρχουν τόκοι που πρέπει να πληρωθούν. Το transfer λοιπόν αυτό προτείνω να γίνει, εγώ λέω να γίνει η μεταβίβαση αυτή, αλλά θα χρειαστούν 10 δισεκατομμύρια ευρώ που προβλέπονται για να καλύψουν τις πληρωμές του 2013. Αυτό σημαίνει ότι παρά την πρώτη αυτή δόση 7,3 δις, του δεύτερου διορθωτικού προπολογισμού που είναι 60% των αγκών του προγράμματος θα λείψουν ήδη για την γραμμή αυτή του προπολογισμού οι πόροι για να φτάσουμε στο τέλος του έτους. Έχουμε το προπολογισμό 17 που βγάζει ε, ε, αποθεματικά από τον προπολογισμό για το λεγόμενο πακέτο που θα θυμάται η κυρία Χορμάγερ είχαμε ορίσει ως πακέτο αποθεματικού Σέγγεν 97,8 εκατομμύρια ευρώ σε δεσμεύσεις και 55,2 σε πληρωμές. Στις 29 Μαΐου επήλθε συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου Κοινοβουλίου για το νομοθετικό πακέτο Σέγγεν, άρα πιστεύω ότι δεν άκουσα και τους συναδέλφους από την ε, ΛΥΜΠΕ. Πιστεύω ωστόσο ότι υπάρχουν, πληρούνται οι προϋποθέσεις για να απελευθερωθεί το αποθεματικό του Σέγγεν. Καλώ τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν λοιπόν την ε, ε την μεταφορά του προϋπολογισμού 17. Προϋπολογισμός 18. Ανθρωπιστική βοήθεια που θα πρέπει να αφορά τη Συρία για 247,7 εκατομμύρια ευρώ δεσμεύσεων και 140 εκατομμύρια πληρωμών. Και εδώ η μεγάλη απουσία των προπολογισμών για τη γραμμή αυτή δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων ρευστότητα. Και επειδή μιλάμε για ανθρωπιστική βοήθεια, ε, Μα ζητούσαν οι συνάδελφοι και από την Προεδρία και από την Επιτροπή Ανάπτυξης να παρέμβουμε υπέρ αυτής της μεταφοράς. Με έγκριση πρώτης δόσης από τις δύο, τις δύο εφόσον θα έχουμε πόρους για να αντιμετωπίσουμε τις πρώτες επίκουσες καταστάσεις. Η ανάγκη ωστόσο, οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες. Επ, αυτού του, επ αυτής της μεταφοράς πρέπει να τονίσω ότι πόροι πρέπει να αντληθούν από ορισμένα προγράμματα προτεραιότητας για το Κοινοβούλιο όπως ε, η ανάπτυξη, η αναπτυξία βοήθεια προς Λατινική Αμερική και Ασία. Αλλά για το σκοπό της μεταφοράς που είναι η υποστήριξη ε, της ανθρωπιστικής βοήθειας θα πρέπει να απελευθερωθεί, να επιτραπεί η μεταφορά και μετά θα δούμε ε, πώς θα χρησιμοποιηθούν άλλοι πόλεις στην Ολομέλεια. Και η παριθμόν 19 μεταφορά για την ανθρωπιστική βοήθεια 15 δεσμεύσεις 8 εκατομμύρια ευρώ πληρωμές για βοήθεια στο Κονγκό και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Και εδώ πιστεύω ότι για ανθρωπιστικούς λόγους για τους οποίους ε, απευθύνονται οι πόροι, θα είναι σκόπιμο να δώσουμε το OK για τη μεταφορά. Μεταφορά 21 που αφορά μόνο πληρωμές και όχι υποχρεώσει, 21 εκατομμύρια ευρώ για το εργαλείο σταθεροποίησης. Λόγω της έλλειψης πληρωμών που οφείλεται στο χαμηλό επίπεδο προβλέπει ο προπολογισμό του 2013. Επρόκειτο για 42 εκατομμύρια ευρώ λιγότερο σε σχέση με αυτό που είχε προβλέψει η Επιτροπή στο σχέδιο προπολογισμού. Είναι σαφές λοιπόν ότι με όλες αυτές τις μεταφορές που προτείνω να υπερψηφίσουμε σήμερα το απόγευμα θα προσπαθήσουμε απλά να βάλουμε κομματάκια κομματάκια υφάσματο σε ένα ρούχο μπαλώματα δηλαδή σε ένα ρούχο που έχει του κόσμου τις τρύπε. Πρόκειται για πολύ μικρή προσπάθεια. Πρέπει να το κάνουμε για να υλοποιήσουμε τα προγράμματα και την, την ανθρωπιστική βοήθεια που είναι ουσιαστικές για πληθυσμό που πλήττονται από προβλήματα όπως την κατάσταση στην Συρία, την, Αφρικανική, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και το Κονγκό. Αυτή είναι η κατάσταση Αυτό πρέπει να ψηφίσουν το απόγευμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και εγώ θεωρώ ότι σήμερα το απόγευμα, α, όταν θα ψηφίσουμε, ότι θα είναι θετική η ψηφοφορία. Πολύ λίγο χρόνο τώρα, ο Φερνάντο. Όχι, συγγνώμη, ο Ζωσέ Μανουέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι λακωνικός. Μία διαπίστωση για το Ταμείο ελληνική. Θα πρέπει να ενεργοποιείται πολύ πιο γρήγορα. η πρόταση για τη Σλοβενία και την, Κροατία και την Αυστρία για τις πλημμύρες ε, ε, έχει ήδη καθυστερήσει γιατί Πρόκειται για περιστατικά Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του 2012. Λυπούμε για την μεγάλη καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης. Άλλωστε προβλέπεται στο διορθωτικό κανονισμό ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης έχει μέχρι και ένα δις ε, ετησίως. Και εδώ μιλούμε για 14.600.000 ευρώ για τους πλημμυροπαθείς στις τρεις χώρες. Πληρούνται άλλωστε οι προϋποθέσεις. Η Σλοβενία έπληγε περισσότερο σε ό,τι αφορά το ποσοστό του ΑΕΠ 0,6% του εθνικού ΑΕΠ ήταν οι ζημιές. Έχουμε 214 εκατομμύρια το κατόφλι και επιπλέον σε αυτό το κατόφλι το όριο επιβάλλεται το ποστό του 6% και το 2,5% για την Κροατία και την Αυστρία. Δεν έχουν φτάσει ε, το 6 του ΕΠ. Βέβαια ήταν μεγάλες οι ζημιές ε, στο 2012 γιατί και αυτές οι δύο χώρες πήγησαν από τις πλημμύρες, οπότε θα πρέπει και αυτές να καλυφθούν από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Τώρα, το περιθώριο λιγμών ήταν 14,8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είχε προβλεφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κινητοποίηση του Ταμείου ε, Αλληλεγγύης εμπίπτει στη δημοσιονομική γραμμή 3β του δημοσιονομικού πλαισίου. Τώρα, επαναλαμβάνω, το ποσό αυτό είναι σχετικά μικρό. Θα πρέπει λοιπόν να μην καθυστερήσει η κινητοποίησή του. Και επαναλαμβάνω, για το Ταμείο Ελεγγύης θα πρέπει να δρούμε πιο γρήγορα, ώστε να κινητοποιείται άμεσα και να είναι έτσι πολύ πιο αποτελεσματικό. Γιατί δυστυχώς παραπονιούνται οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, για τις καθυστερήσεις, κάτι που αμαυρώνει την ε, εικόνα του Ταμείου Αλληλεγγύης. Ιδιαίτερες εθεομηνίες θα πρέπει να κινητοποιείται πολύ πιο γρήγορα για να ελαφρύνονται οι ζημίες από τέτοιες εθεομηνίες. Ευχαριστώ πρωτού συμπληρώσει, μάλλον δώσει, να δώσω το λόγο στον Τζιωβάνι να συμπληρώσει, αλλά πρώτα να ακούσουμε και του υπόλοιπου ε, ομιλητέ. Έτοιμα ήταν, δεν ήταν πρόταση, έτοιμα προς την Προεδρία για το σημείο 19 της με Διάταξης βατικά μέτρα για την ανάπτυξη της Πένθου, για την κοινή γεωργική πολιτική. Να μην συζητηθεί αυτό το απόγευμα, διότι η ψηφοφορία στην Επιτροπή Γεωργίας θα γίνει τέλη Σεπτεμβρίου, οπότε έχουμε άνετα τη δυνατότητα να το δούμε Σεπτέμβριο όταν θα έχουμε και την έκθεση της Επιτροπής ε, Γεωργίας. Μάλιστα, θα το διαγράψουμε λοιπόν από την ημερήσια διάταξη αυτό. Έντα και οι διερμηνείς μας δίνουν πέντε λεπτά ακόμα, αν θέλετε, αν έχετε την καλοσύνη. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι λακωνική. Έχω μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το δεύτερο τμήμα του δεύτερου διορθωτικού προπολογισμού, Γιατί ήδη το Συμβούλιο έχει εγκρίνει το πρώτο τμήμα του υπαριθμού 2 διορθωτικού προπολογισμού και έχει ε, προταθεί συμβαστική λύση για το δεύτερο τμήμα. Αλλά φαντάζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρειαστεί να υποβάλει δεύτερο διορθωτικό προπολογισμό που να περιλαμβάνει το δεύτερο τμήμα και ίσω και κάτι επιπλέον. Διπλή λοιπόν η ερώτηση. Πότε θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το διορθωτικό προπολογισμό. και Ποιο πιστεύετε θα είναι το ποσό αυτού του διορθωτικού προπολογισμού υπαριθμών 2. Και τώρα για τις μεταφορές που μας παρουσίασε ο Τζοβάνι Λαβία. Έχουμε πέντε μεταφορές πιστώσεων που θα πρέπει να ψηφίσουμε το απόγευμα. Και φυσικά θα υπερψηφίσουμε. Τέσσερις από τις μεταφορές αυτές οφείλονται σε προβλήματα πληρωμών ή σε μη έγκαιρη ε, έγκριση ε, και εμπρόθεσμη ε, έγκριση του διορθωτικού προπολογισμού λόγω εξαιτία του Συμβουλίου ή γιατί δεν είχαν προβλεφθεί στον προπολογισμό το 2013 αρκετά πιστώσει πληρωμών. Και ήδη στο παρελθόν είχαμε πει ότι δεν μας φτάνουν ε, οι πληρωμές και αυτό δεν το λέγαμε για να ενοχλήσουμε το Συμβούλιο είτε για να το πιέσουμε. Ιδού η απόδειξη. Είχαμε δίκιο δικαιολογημένα ζητούσαμε περισσότερες πιστώσεις πληρωμών με βάση τα στοιχεία που είχαμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάστηκε τώρα διορθωτικός προϋπολογισμός. Και πολύ σημαντικό θέμα που λαμβάνουμε εμείς υπόψη και όχι το Συμβούλιο είναι οι συνέπειες ε, της ε, μη εμπρόθεσμης καταβολής των πληρωμών. Πρόστιμα, υπερημερίες, ε, προβλήματα για τις επιχειρήσεις και ακόμη πιο αρνητικές συνέπειες για την ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν θα πρέπει να μας ξεχάσετε πάλι στις διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν όσον για τον προϋπολογισμό του 2013 με όλους τους ασφικτικούς κλειούς που μας επιβάλλει το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο κύριος Πλένκοβιτς. Ε, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στην έκθεση στις έκθεσεις που έχουν να κάνουν με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να αναφερθώ στις καταστροφικές συνέπειες των ε, όσων συνέβησαν στην Σλοβενία, την Κροατία, την Αυστρία. Σε ό,τι αφορά την Κροατία, πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ και αυτό επηρεάζει εννέα κομιτείες της ε, Κροατίας και ε, πραγματικά αυτό επηρέασε 800.000 άτομα και τις ζωές τους. Ήταν πραγματικά βαθύς ο αντικτύπος. Ήταν η δεύτερη περίπτωση όπου χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί το Ταμείο Αντιλεγγύης στην Κροατία λόγω των περιστατικών το 2010 και το 2011. 14,6 εκατομμύρια ευρώ σκοπεύει να κινητοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάνω από 14 θα ε, χρησιμοποιηθούν για την Σλοβενία και για την Αυστρία και την Κροατία θα είναι πολύ πιο μικρό το ποσό. Αλλά επειδή είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε αυτό στην Ευρωπαϊκή, στην Επιτροπή Προπολογισμών, υπάρχει δυνατότητα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κονδύλια αυτά για την Κροατία να αυξηθούν. Δεν ξέρω αν ο κύριος Πρέζα επιθυμεί να απαντήσει. Thank uh, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να απαντήσω συντομία στο ερώτημα που έθεσε ο κύριος η κυρία Κατασάμπα για τις μεταφορές αυτές. απαντήσω ότι από ό,τι φαίνεται το προπολογισμό είναι επαρκή όπως έχει δημορφωθεί και στον τροποποιημένο προπολογισμό υπαριθμό 2 δεν έχουν ακόμα γίνει συγκεκριμένες προτάσεις. Άρα, για να ανταποκριθούμε στις πιο άμεσες ε, ανάγκες, όπως είπε ο κ. Λαβία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί προσπαθεί να μεταφέρει τέτοιες ε, πιστώσεις πληρωμών από το ένα μέρος στο άλλο για να σβήσει τις πιο κατεπίγουσες φωτιές αν θέλετε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσβλέπει στην έγκριση του τροποποιημένου προϋπολογισμού της κατηγορίας 2 που είναι η πιο επίγουσα. Στην παρούσα φάση ο διευθυντικός προϋπολογισμός υπαριθμών 2 που ε, προαπαιτεί 11,2 δισεκατομμύρια εξακολουθεί να υφίσταται, έχει τροποποιηθεί από το Συμβούλιο και θα εγκριθεί κατά πάσα πιθανότητα το Σεπτέμβριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν το χρόνο θα παρουσιάσει την, ε, τις υπόλοιπες δόσεις, την, απομείνουσα δόση και ενδεχομένως να χρειαστεί να αναθεωρήσει την κατανομή μεταξύ των διαφόρων ε, σημείων του προπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταφορές που έχουν προσωρινή φύση για να ανταποκριθούν στις πιο κατεπίγουσες ανάγκες. Να σας πω όμως ότι και τα 11,2 δισεκατομμύρια ευρώ χρειάζονται. Αυτό πέρα από κάθε αμφιβολία δεν υπάρχει περίπτωση θα χρειαστούν, να χρειαστούν λιγότερα χρήματα. Για το ερώτημα του κ. Μπρανκοβίτς, για το νέο ταμείο, για, για νέο ταμείο αλληλεγγύης για την Κροατία έχουν εκτιμηθεί τα ποσά εφαρμόζοντας τους κανόνες επιλεξιμότητας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης και τα σχετικά ποσά θα προσαρμοστούν στην... με την πάρδα του χρόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η κυρία Γιούτα Ευχαριστώ και πάρα πολύ τους ε, διερμηνείς που έμειναν μαζί μας ε, πιο πολύ ώρα από ό,τι προβλεπόταν. Να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους αλλά και στους ε, σε καλή όρεξη. Οι, συντονιστές στις, οι συντονιστές στις 2. Θα τα ξαναπούμε στις δύο με τους συντονιστές.